Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Έχουμε την ημερήσια διάταξή μα σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο. Υπάρχουν αντιρρήσει σε ό,τι αφορά την ημερήσια διάταξη. Εάν όχι, θεωρούμε πω εκρίνεται, χωρί καμία αλλαγή. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 19η και 20η Νοεμβρίου, τη 3η Δεκεμβρίου και τη 10η Δεκεμβρίου. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις κάτι διάρκεια τη συνεδρίασής μας ε, σήμερα από την πλευρά σας θα θεωρηθούμε πως εγκρίνονται και αυτά τα πρακτικά. Σημείο 3. Οι ανακοινώσει ε, που έλαβαν οι συντονιστέ κατά τη συνεδρίασή του στι 19 Νοεμβρίου έχουν συμπεριληφθεί στα πρακτικά ε, τη συνεδρίαση τη Επιτροπή και εν λόγω αποφάσεις, οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και αν δεν εκφραστούν αντιρρήσεις στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, θεωρούμε πως εγκρίνονται και αυτές οι αποφάσεις. Σημείο 4. Να σας ενημερώσω ότι ο συνήθως ε, η εν λόγω συνεδρίαση ε, είναι web streamed, οπότε από το Λίσαβονο στο Λούνεμπουργκ και από το Ταλίνο στη Θεσσαλονίκη καλωσορίζω όλους τους τηλεθεατές μας. Και καθώς υπάρχει διερμηνία σήμερα, σας παρακαλώ να μιλάτε δυνατά, καθαρά και όχι πολύ γρήγορα. Και σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ, έχει οριστεί για τις 8 Φεβρουαρίου στις 6. Και αυτό οφείλεται στην ε, καθυστερημένη εξέταση της εν λόγω Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου από την πλευρά του Συμβουλίου. Θα δούμε από εδώ και πέρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ε, μέχρι στιγμής θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουμε στο πλαίσιο δηλαδή του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος να κρίνουμε την Ελληνική συμφωνία. Θα δούμε όμως. Σημείο 5 τώρα. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και το έχω μαζί μου τον ε, Ζαν Μάτι από την Επιτροπή και να σα ενημερώσω ότι η Σεσίλια Μάλμστρομ ε, βρέθηκε στη Νέα Υόρκη την δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και την τελευταία Παρασκευή η Επιτροπή δημοσίευσε το σχέδιο των δύο διαπραγματευτικών εντολών για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες συνεδρίασε και η ομάδα παρακολούθησης στο Monitoring Group ε, και συζήτησε ε, περισσότερο σε βάθος την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων και είναι ξεκάθαρο πως σε αυτή τη χρονική συγκυρία υπάρχει μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τη σχέση που έχουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Το ζητούμενο είναι από τη μία πλευρά να επιτύχουμε μια αποκλιμάκωση και από την άλλη πλευρά βέβαια να επιμείνουμε στις δικές μας προτεραιότητες. και απο την αλλη πλευρα βεβαια να επιμεινουμε στις δικες μας προτεραιοτητες ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η Επιτροπή και ο Ζαν Λουκ θα μας εξηγήσει ε, τώρα τι ακριβώς κάνει η Επιτροπή από την πλευρά τη. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα παραμείνουν υψηλή προτεραιότητα στου επόμενου μήνε. Θα συνεχίσουμε τις επαφές μας με την Αμερικανική Διοίκηση σχετικά με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ακόμα και κατά στενών εταίρων. Υπάρχουν κάποιες εντάσεις μεταξύ του Προέδρου και του Κοινοβουλίου και υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις αμερικανικής νομοθεσία υπό τι οποίε θα μπορούσε να έχει ένα περιθώριο λιγμών ο πρόεδρο. Εμείς θα πρέπει να διατηρήσουμε την ηρεμία μας και η προτεραιότητά μα παραμένει να υλοποιήσουμε όλες τις πτυχές της κοινή δήλωσης της 25ης Ιουλίου. Θα πρέπει να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τα όσα συμφωνήσαμε και μιλώ μόνο για το joint statement. Θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και την, τον εξυγχρονισμό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από κρατικού τύπου καπιταλισμό, λέει ο μιλητής. Στον ΠΟΕ υπάρχει σημαντικός κίνδυνος το σώμα προσφυγών να μην είναι πλέον επιχειρησιακά έτοιμο λειτουργικό. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε έναντι οποιοδήποτε μέτρου κατά του ελεύθερου εμπορίου θα μπορούσε να αναλυφθεί από την Αμερικανική διοίκηση. Και μιλώ για ποσοστώσεις για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και ανταλλακτικά. Εμείς εκεί θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές ότι είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε θα μπορούσαμε να λάβουμε αντισταθμιστικά κέντρα επί συνολικής αξίας ε, εμπορεύματα 20 δισεκατομμυρίων και για τα οποία οι Αμερικανοί δεν είναι ο κυρίαρχος προμηθευτής. Εφόσον όλα αυτά απαιτηθεί η κατάσταση είναι τέτοια κατά την οποία θα πρέπει να αναλάβουμε μέτρα. Σύμφωνα πάντως με τις συμφωνίες μεταξύ των δύο προέδρων τον Ιούλιο θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια να έχουμε ένα θετικό θεματολόγιο εμπορικό και επί της ουσίας και προκειμένου να μην πάμε σε πολύ αρνητικές σε καταστροφικών συνεπειών θέσεις αναδίπλωσης. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ευκταίο να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε πλήρη εμπορική συμφωνία με την Αμερικανική πλευρά. Και δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουμε σε διαπραγματεύσεις τύπου TTIP. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Η διαπραγμάτευση TTIP απέτυχε. και καλό είναι να μην επιβαρύνουμε, επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο τα πράγματα εκεί. Την, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε δύο σχέδια οδηγιών για δασμολογικές ποσοστώσεις και έχουμε και αξιολογήσεις ε, συμμόρφωση. Αυτό είναι αρκετά περίπλοκο θέμα. Ισοδυναμίας μάλλον, ώστε να είμαστε σίγουροι για τη θέση σε εμπορία συγκεκριμένων προϊόντων που καλύπτουν όλα τα πρότυπα ή αντίστροφα ώστε τα προϊόντα που δεν καλύπτουν πρότυπα ασφαλείας να μην μπορούν να τίθεται σε εμπορία. Έχουμε όμως αποκλήσεις προσέγγισης σε αυτές τις ε, αξιολογήσεις ε, ισοδυναμίας, συμμόρφωσης στην ουσία, χωρίς όλα αυτά να οδηγούν σε αυξημένη ασφάλεια για τα προϊόντα. Η δική μας σύσταση είναι να μειώσουμε το περιττό κόστος διατηρώντας το ίδιο επίπεδο προστασίας δεν πρόκειται όμως για διαπραγμάτευση επί των δικών μας προτύπων ή του δικού μας επίπεδου προστασίας. Έχουμε διακριτά σχέδια επί των οποίων θα μπορούσε να σημειωθεί επιμέρους πρόοδος με τη διακυβέρνηση Τραμπ και στα, στο πεδίο των ιατροφαρμακευτικών η Κομισιόν έχει διαπραγματευτική εντολή και ίσως να, μπορούμε, να, να μπορέσουμε να έχουμε θετικές ε, επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές επαναλαμβάνω σε επιμέρους συμφωνίες. Σε καμία περίπτωση όμως ε, δεν θα θέλαμε να προτείνουμε την έναρξη διαπραγματεύσεων ε, ε, συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών για δημόσιες προμήθειες, θαλάσσιες υπηρεσίες, γεωγραφικούς προορισμούς, SPS. Γιατί κατέστη αδύνατον για τους Αμερικανούς να κινηθούν ακόμα και ένα χιλιοστό σε αυτά τα παιδιά Και το οποίο οδήγησε στην ουσία και στην ε, αποτυχία των διαπραγματεύσεων TTIP ε, στο τέλος του 2016. Και ένα από τα βασικότερα διδάγματα της TTIP είναι ότι <clears throat> το ρυθμιστικό θεματολόγιο με τους Αμερικανούς καλύτερα να το αναπτύσσουμε εκτός του κλασικού πεδίου FTA. Πρέπει λοιπόν, επαναλαμβάνω, να κοιτούμε επιμέρους σημεία στα οποία μπορούμε να σημειώσουμε μικρή πρόοδο, αντί να κοιτούμε ευρύτερα πλαίσια. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά την ε, κατάσταση και προσβλέπουμε στην περαιτέρω συζήτηση μαζί σας. Είμαι έτοιμος να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση. first I will give the floor to the standing... Να δώσω το λόγο στο μόνιμο εισήγητη για τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και μετά στους Σκιώδης. Λοιπόν, αλλάζω καπέλο και είμαι ο εισηγητής σας πλέον για τα θέματα των εμπορικών σχέσεων σε ένα σημείο θα συμφωνήσω απόλυτα με την παρουσίασή σας. Δεν είναι δυνατόν κάτω από τις παρούσες συνθήκες να διαπραγματευτούμε μια συνολική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, ε, υπό την κυβέρνηση αυτή τουλάχιστον. Ίσως και ανεξαρτήτως της κυβέρνησης που έχει την εξουσία στην Ουάσιγκτον. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και σε σχέση με τις δημόσιες προμήθειες και σε σχέση με τις υπηρεσίες και τα εργασιακά δικαιώματα και τα λοιπά. Συνεπώς λοιπόν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Και αυτή είναι και η εμπειρία που ζήσαμε με το TTIP. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε μήπως μπορούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις σε μια διαφορετική βάση και έχω εδώ κάποιες ερωτήσεις. Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν υποπίεση. Έχουμε στοιχεία πίεση στην παρούσα φάση. Καταρχάς, οι δεσμοί ε, στον τομέα του αλουμινίου και του χάλιβα εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. Και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών από ό,τι λένε ε, για να τερματίσουν τους δεσμούς αυτούς. Και δεύτερον, έχουμε τις απειλές για δασμολογικά μέτρα στην αυτοκινητοβιομηχανία και τα ανταλλακτικά. Υπάρχει δηλαδή πάντα ο κίνδυνος, υπάρχει η απειλή, εν πάση περιπτώσει, επιβολής δασμών στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων τα οποία προέρχονται από ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Και όλα αυτά ήταν βέβαια τμήμα των διαπραγματεύσεων στο παρελθόν. Το θέμα είναι, τίθενται δύο ερωτηματικά για τις δύο αυτές απειλές. Καταρχάς, σε ποιο βαθμό έχουμε διαφορές με τις προηγούμενες, είναι σαφείς οι διαφορές με τις προηγούμενες καταστάσεις τον Ιούλιο υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία λέγοντας ότι δεν ε, θα δεχθούμε για δίποτε συμφωνία χωρίς αναφορά στην ε, Σύμβαση των Παρισίων για το κλίμα. Οπότε στην παρούσα φάση ε, η απόκριση από πλευράς των ΗΠΑ γνωρίζουμε ποια είναι. Ταυτόχρονα όταν συζητάμε εμπορικές συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕ και των ΚΑΤΟ παλαιών, λέμε ότι θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο γενικά των εμπορικών δραστηριοτήτων. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι μιλάμε μόνο για βιομηχανικά είδη εκτός αυτοκινήτων, κάτι το οποίο δεν είναι αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε και δεν καλύπτονται όλα αυτά τα οποία θα είχε ζητήσει να, να συζητηθούν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε και άλλες διαφορές, όπως σαν παράδειγμα το ε, διαιτητικό ή εφετικό σώμα και διαρωτώ με αν υπάρχει ε, κάποιο μήνυμα από πλευρά των ΗΠΑ ότι αν αρχίσουν διαπραγματεύσεις εκ νέου θα μπορούσαν να αλλάξουν τη θέση τους γύρω από αυτό. Λοιπόν, αυτός, αυτές ήταν οι ερωτήσεις προς ε, τον κύριο Ντεμαρτή και τώρα δίνω το λόγο στην πρώτη σκιώδη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να θυμάστε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Χαίρομαι για την παρουσία σας εδώ. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε. Αλλά αν πράγματι προσπαθούμε να αποτρέψουμε τον οικονομικό πόλεμο με τις Ηνωμένε Πολιτείες, και να αποφύγουμε τις ζημίες από μια πιθανή επιβολή δασμολογικών κυρώσεων, θα πρέπει να ορίσουμε σωστά τα θέματα τα οποία επιλέγουμε προς συζήτηση και στα οποία θα είχαμε κάποιες δυνατότητες επιτυχίας. Ή μήπω δεν θα έπρεπε να μπούμε καθόλου σε διαπραγματεύσεις. Αν ορίσουμε ένα τμήμα προς διαπραγμάτευση αυτό μπορούσε να αποτελέσει ένα κίνδυνο για το σύνολο των σημείων τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δεμαρτή για την ενημέρωση την οποία μας έκανε σε σχέση με τις επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ. Και πράγματι είναι σαφής η επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πάρει την εντολή του Συμβουλίου έτσι ώστε να ξεκινήσει ε, την διαπραγμάτευση αυτή και ε, με τις ε, ερωτήσεις τις πέντε τις οποίες σας έθεσε ο Πρόεδρός μας συμφωνώ. Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ο κίνδυνος πιθανότητας επιβολής υπερεδαφικών κυρώσεων σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις τις οποίες διατηρούμε με τρίτες χώρες. Αυτό πώς ε, επηρεάζει τις συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις ε, για τα αγαθά και τα εμπορικά προϊόντα και σε ποιο βαθμό θα χαρακτηρίσει τις συζητήσεις που επιθυμείτε να ξεκινήσετε. Αναφερθήκατε ήδη στην νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών τη λεγόμενη 232 σε ποιο βαθμό αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια απειλή για κάποιες κατηγορίες προϊόντων οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τις εμπορικές μας δραστηριότητες. Σε ποιο βαθμό δηλαδή οι ρυθμίσεις του 3 του απειλούν αυτές τις δραστηριότητες. Ε, θα ήθελα να μας πείτε επίσης ε, για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε διοικητικό επίπεδο για το χάλιβα και το αλουμίνιο, αλλά το του, είναι θα έλεγα νομική ρύθμιση. Και σε ποιο βαθμό μια τέτοια νομική ρύθμιση μπορεί να ανακληθεί έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία. Γιατί στην παρούσα φάση η ρύθμιση αυτή αποτελεί ένα νομικό περιορισμό Πώς εσείς θα θέσετε το θέμα αυτό ε, στα υποδιαπραγμάτευση θέματα. Ξέρω ότι έγιναν και άλλες συζητήσεις μέχρι τώρα. Ξέρω ότι τα αγροτικά προϊόντα, σαν παράδειγμα, έχουν εξαιρεθεί. Ενώ από την άλλη ακούμε βέβαια από πλευρά των ΗΠΑ ότι επιθυμούν τη συζήτηση και για τα γεωργικά προϊόντα. Τι ακριβώς θα τεθεί λοιπόν υπό συζήτηση. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι τα αγροτικά δεν θα τεθούν προς συζήτηση. Σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων. Η φωνή σας έχει αλλάξει λίγο. Μου θυμήσατε λίγο τη φωνή της Ζάρα Λέαντα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αν θυμάμαι τις δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει από πλευρά της Επιτροπής στο παρελθόν, η διαπραγμάτευση με τη ΣΥΠΑ στο συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο είναι συζητήσεις με το πιστόλι στον κρόταφο. Δεν ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να αλλάξει την εντολή διαπραγμάτευσης με τους Αμερικανούς, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ε, το πιστόλι αυτό εξακολουθεί να είναι γεμάτο και απειλητικό. Πήραμε κάποιες διαβεβαιώσεις σχετικά με την εξαίρεση της Γεωργίας από τα προσδιαπραγμάτευση θέματα, αλλά έχω ανησυχίες γι' αυτό, γιατί βλέπω ότι ε, το, η Αμερικανική Γερουσία συνεχίζει να λαμβάνει μέτρα περιορισμού εισαγωγής ευρωπαϊκών προϊόντων και γνωρίζουμε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν οι Αμερικανοί έτσι ώστε τα προϊόντα τους, τα γενετικά τροποποιημένα και τα κρέατα τους, τα βοηδή γεμάτα ορμόνες θα πλημμυρίσουν κάποια στιγμή την ευρωπαϊκή αγορά. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τη Γερμανία η οποία φοβάται τις περιορισμούς στις εξαγωγές. Ε, το θέμα είναι να προσπαθήσουμε η Γεωργία να παραμείνει εκτός διαπραγματεύσεων και μετά από την εντολή του Συμβουλίου. Αυτό θα πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύν της άλλης ε, και για τις πιθανές απειλές των τομέα ρύθμισης ε, των και εποπτείας των ερευνών και των δοκιμών νέων φαρμακευτικών προϊόντων και ουσιών. Ξέρουμε τι απειλούν οι Αμερικανοί και στον συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία τίθενται υπό αμφισβήτηση. Συνεπώς λοιπόν δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε αδίποτε μορφή συμφωνίας η οποία να θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και συγκεκριμένους τομείς βιομηχανικούς έτσι ώστε ένα νέο TTP να μην γίνει ποτέ πραγματικότητα. Σέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Λάγκα. Να πω ότι κατά τη δική μου άποψη το σημείο αφετηρίας είναι ότι ναι, είναι θετικό το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε διάλογο και ότι έχουμε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση. Γιατί το πρώτο βήμα είναι να βρεθούμε στην ίδια αίθουσα και να αρχίσουμε να ε, μιλάμε μεταξύ μας έτσι ώστε να αποφύγουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Άρα λοιπόν αυτό είναι θετικό. Από την άλλη όμως ε, πλευρά θεωρώ πως ε, είναι η κατάλληλη στιγμή για να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα και να μετριάσουμε τις προσδοκίες μας. Και ίσως ακριβώς αυτό το μετριασμό των προσδοκιών θα πρέπει να τον είχαμε εφαρμόσει κατά την προετοιμασία της συμφωνίας TTIP. Δηλαδή, αυτέ οι διαπραγματεύσει που έχουμε ξεκινήσει δεν μπορούν να επιλύσουν τα, τα πάντα, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση σε επίπεδο ΠΟΕ, σε ό,τι αφορά ε, το πρόβλημα της ε, συμφωνία με το Ιράν ε, και ένα σωρό περαιτέρω ζητήματα. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα πάντα. Και για να είμαι και πιο ειλικρινή, μπορούμε τελικά να επιτύχουμε μια βασική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ακόμα και αυτό δηλαδή τίθεται να αμφιβόλω σε κάθε περίπτωση για να επιτύχει κανείς ε, μια συμφωνία καταρχήν θα πρέπει να ορίσει το αντικείμενο αυτής της συμφωνίας ε, και διαβάζοντας τα διαφορετικά έγγραφα, το έγγραφο της δικής μας εντολής, ε, το κείμενο από την πλευρά των Αμερικανών βλέπω ότι τελικά οι προσδοκίε ω προ το τι θα συζητηθεί είναι εντελώ διαφορετικέ. Από τη μία ε, πλευρά ε, λέμε ότι δεν θέλουμε να υπάρξει συμφωνία TTIP, αλλά τελικά εμεί επιθυμούμε το ίμιση, αν θέλετε, των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε μια συμφωνία TTIP και οι Αμερικανοί θέλουν το άλλο ίμιση των όσων θα περιλαμβάνονταν σε μια συμφωνία ε, TTIP. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα αντικείμενα εκείνα τα οποία θέλουμε εμεί να συζητήσουμε και ποια είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν εκείνοι. ε, αντιλαμβάνομαι την ε, πολιτική συγκυρία, το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή το πολιτικό, ε, το οποίο μας οδηγεί στο να θέλουμε να έχουμε μια στενή, αν θέλετε, διαπραγματευτική εντολή, δηλαδή μια περιορισμένη εντολή. Από την άλλη πλευρά όμως θέλουμε οι συμφωνίες τις οποίες συνάπτουμε να είναι ευρείες, γιατί κάτι τέτοιο είναι ε, προς ε, όφελός μας. Αλλά από την άλλη πλευρά θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα και δικά μας επιθετικά συμφέροντα, offensive interests, Μόνο Αμερικανοί έχουν. Πάντω, σε κάθε περίπτωση, εγώ να πω πω η εντολή για την TTIP ε, μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μα επέτρεπε να προβούμε στη διαπραγμάτευση ε, μια ευρεία συμφωνία. Τι έχει συμβεί όμω τώρα με, αυτή, εκείνη την εντολή, δηλαδή δεν ισχύει πλέον, είναι νεκρό γράμμα, είναι λόγω εντολή για την ε, TTIP ή έχουμε δύο διαφορετικές εντολές σε ό,τι αφορά δηλαδή το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων όπως αυτό θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Πέντε ακόμα ομιλητέ έχουν ζητήσει το λόγο και κλείνω εδώ τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρε, και ευχαριστώ, κύριε Ντεμάτη. Θα επανέλθω σε κάτι που ε, αναφέρατε ε, στην αρχή της παρέμβασής σας ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και συνεπής. Ε, και αυτό πράγματι αυτή τη στάση θα πρέπει να την τηρήσουμε έναντι κάποιου ο οποίο είναι πολύ πιο ασταθής ε, επιθετικό. Αλλά νομίζω πω η αίσθηση που δίνουμε στο ευρύ κοινό είναι ότι η τακτική έτσι, εκφοβισμού που ακολουθεί ο πρόεδρος Τραμπ ε, αποφέρει καρπούς γιατί μας αναγκάζει δηλαδή να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οπότε αυτό είναι σημαντικό από άποψη ε, ε, εντύπωση στην οποία δίνουμε προς τα έξω. Γιατί βέβαια γνωρίζουμε και στο επίπεδο της εξωτερικής ε, πολιτικής υπάρχει αυτή η συνιστόσα του ποια είναι η αίσθηση δίνουμε προς τα έξω. Πάντως θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο συνάδελφος ότι δηλαδή εν ώψη ενός εθνικού εμπορικού πολέμου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μείνουμε σε διάλογο και να έχουμε όλες τις δυνατότητες ανοιχτές. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Αν δούμε πόσο είχαν προχωρήσει οι διαπραγματεύσει σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στοιχεία τη TTIP, γιατί γνωρίζω πω υπάρχουν άλλα στοιχεία στα οποία πραγματικά βρισκόμαστε σε αντίεξοδο. Για παράδειγμα, όμω, σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά αγαθά, είχαμε προχωρήσει αρκετά σε διάφορε ομάδε εργασία σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση. Οπότε το ερώτημά μου είναι το εξή. Υπάρχει ήδη ένα κομμάτι εκείνων των εργασιών το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για την περαιτέρω διαπραγμάτευση ε, και θα τύχει βασμό από την Αμερικανική πλευρά όλο αυτό το κομμάτι το οποίο είχαμε δηλαδή ε, καταλήξει σε προσωρινές συμφωνές. Γιατί με βάση τι εντολέ που υπάρχουν σήμερα νομίζω πως ε, πράγματι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε γρήγορη διαπραγμάτευση βασιζόμενα στα όσα ήδη είχαμε συζητήσει στο πλαίσιο τη προετοιμασία τη TTIP. Δεύτερο ερώτημα τώρα λαμβάνοντας υπόψη μας ε, το, την κλίμακα εδώ του μερους εμπορίου, ουσιαστικά στην ουσία πρόκειται για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και στη στρατηγική της ε, εμπόριο για όλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες η βιώσιμη ανάπτυξη θα αποτελέσει στοιχείο κλειδί. Και βέβαια σε σχέση με τις ΗΠΑ βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ε, κατάσταση, γιατί σε ό,τι αφορά το βιομηχανικό τομέα και το τομέα της μεταποίησης υπάρχει ένα κοινωνικό ντάμπινγκ το οποίο λαμβάνει η χώρα ε, ειδικότερα λόγω της ε, παραβίασης των προτύπων σε ό,τι αφορά την εργασία από, τα, από τις πολιτείες του Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι παραδοσιακά ισχύουσες συνοδευτικέ συμφωνίε που υπάρχουν στον τομέα τη εργασία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτω ώστε να δούμε τι ακριβώ θα συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, ο κύριο Μπούχνερ. Ναι, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η διαφάνεια και πώ θα την εξασφαλίσουμε. Δηλαδή, ε, αυτό που έθεσε η κυρία Μπίργκερ, να συμφωνήσω και εγώ ε, με αυτό, ε, ό,τι αφορά το ερώτημα που έθεσε ε, σε σχέση με τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, και τα σχετικά υλικά. Δηλαδή θα αποτελέσουν αυτά τα GMOs ε, αντικείμενο διαπραγμάτευση στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία; ή όχι. Κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, βλέπουμε να έχουμε πολύ διαφορετικέ απόψει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Δηλαδή, στι ΗΠΑ τα δεδομένα είχαμε μεταχείριση ως αγαθό, εμπορικό αγαθό. Βλέπουμε δηλαδή πώς η Google και άλλες επιχειρήσεις διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα. Οπότε ε, ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ήδη ε, υπησέρχεται, αν θέλετε, η αμερικανική νομοθεσία μέσα στην δική μας νομοθεσία προστασία των δεδομένων. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο στο πλαίσιο μιας ε, μελλοντική συμφωνίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ έχω εκπλαγεί από το γεγονός ότι βρίσκεται ε, και πάλι ε, συζήτηση όλο αυτό το κομμάτι της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ αφού ε, δεν είχαμε καταλήξει σε συμφωνία σε ό,τι αφορά την TTIP γιατί ακριβώς η απόψη μας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, ε, την κλιματική αλλαγή και ούτω καθεξής υπήρχαν τεράστιες διαφορές σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Ε, και ε, όλες αυτές οι απειλές τις οποίες ε, έχουμε ακούσει από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ δεν είμαστε επιπισμένοι ότι δεν θα τις υλοποιήσει. Οπότε πώς υπάρχει πρόθεση ξαφνικά από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διαπραγματευτούμε με τον Πρόεδρο Τραμπ. Τι θα κάνουμε δηλαδή και πώς θα σεβαστούμε τις δικές μας αξίες σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα ζητήματα που σας ανέφερα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κλίμα, την προστασία της ε, ε, ε, ευμερίας των ζώων και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή η βασική απέτηση αμοιβαίας, ε, ε, ε, η βασική απέτηση να υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι σε εμά. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Και υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να μου εξηγήσετε πώς αξιολογείτε αυτή την νέα διαπραγματεύση. Επόμενο ομιλητή. Ναι, εμένα με εκπλήσουν λίγο τα αρνητικά σχόλια που ακούστηκαν σήμερα εδώ, γιατί θεωρώ πω οι ε, διαπραγματεύσει θα πρέπει να συνεχιστούν. Οι διαπραγματεύσει σε ό,τι αφορά την TTIP, για παράδειγμα, ε, δεν αβάγησαν ε, <clears throat> επειδή εμεί ήμασταν υπέτειοι, αλλά επειδή η αμερικανική πλευρά δεν ήθελε να προχωρήσει περαιτέρω, να είναι πιο διαλλακτική. Ε, και δεν <clears throat> μπορούμε να ακολουθήσουμε τη λογική ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η μεγαλύτερη χώρα ε, του κόσμου και επιβάλλεται σε όλου. Όχι, ο πρόεδρο Τραμπ και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι μεγαλύτερε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει ε, να ξεκινήσουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει με αυτοπεποίθηση και να γνωρίζουμε ότι ε, εάν δεν επιτρέψουμε στις ΗΠΑ Πολιτείες να διασπάσουν το κοινό μας μέτωπο, τότε είμαστε πιο ισχυρός ε, εταίρος μέσα σε αυτή τη συμφωνία, μέσα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό νομίζω πως θα πρέπει να δώσουμε μια αντίστοιχη εντολή στην Επιτροπή. Είδαμε κατά τους τελευταίους ε, μήνες πως οι προσπάθειες ε, που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ να δημιουργήσει αυτές τις Ε, οι προσπάθειες που έκανε η κυρία ε, Μέρκελ με την επίσκεψή της εκεί αλλά και συνέχεια από την πλευρά του Πρόεδρου Μακρόν όπου πάντα γινόντουσαν οι, ε, οι προσπάθειες από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ να ε, διασπάσει αν θέλετε την κοινή μας γραμμή και το ίδιο ακολούθησε και με την περίπτωση της συνάντησης με τον Ζαν claude Γιούνκερ να πω πως ε, νομίζω πως έγινε αντιληπτό ότι εμείς δεν διασπούμε αυτό το κοινό μας μέτωπο ως Ευρωπαϊκή Ένωση και έκτοτε υπάρχει μια περισσότερη ομαλότητα, περισσότερη ησυχία. Συμφωνώ λοιπόν με όλου του άλλου ομιλητέ ε, που, ε, που είπαν, όπω για παράδειγμα ο συνάδελφο Φιένερ, ότι μπορούμε να είμαστε και λίγο πιο επιθετικοί μέσα σε αυτέ τι διαπραγματεύσει και α δούμε Ε, Πώ ε, μπορούμε για παράδειγμα να ε, υπερασπιστούμε πιο επιθετικά τα δικά μας συμφέροντα γιατί τελικά υπάρχουν και στοχοί, ε, συγγνώμη, τομείς στους οποίους οι Αμερικανοί φοβούνται ότι ενδεχομένω να μην υπάρξει η κατάλληλη ανταγωνιστικότητα από την δική του πλευρά. Και νομίζω πω και στο πλαίσιο των εσωτερικών μα διεργασιών κατά τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, προ τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ενημερώνει το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τέτοιου είδου διαπραγματεύσει και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν νομίζω πω είναι θετικό το να δώσουμε μια τέτοια διαπραγματευτική έντολη ε, στην Επιτροπή. Συνάδελφο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, Πρόεδρε και καταρχήν ε, και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πραγματικά ε, μετά από τόσο ε, μεγάλες ζημιές αν θέλετε ε, το σκαμμένη υγεία των εισαγωγικών βλέπουμε και πάλι να ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Πράγματι το ζητούμενο είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω κλιμακώσεις όπως ε, τις είδαμε στο παρελθόν. Εάν λοιπόν ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση και αν ξεκινήσουμε τους ε, απαραίτητους διαλόγους τότε ενδεχομένως να μπορέσουμε να βρούμε την κατάλληλη άγουσα προς μια εξομάλυνση των σχέσεών μας οι συζητήσεις τις οποίες είχαμε κάνει και εκτός ε, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά ε, τα εμπόδια ε, στο εμπόριο μη δασμολογικού χαρακτήρα θα θυμηθούμε ότι υπήρξαν εδώ κάποια πιο σημαντικά, πιο κρίσιμα στοιχεία σε, αυτή, σε εκείνη τη διαπραγμάτευση και κάποια λιγότερο κρίσιμα. Οπότε ας είμαστε ανοιχτοί στη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσουμε ούτως ώστε να μην υπάρξει μια αρνητική ενημερωτική εκστρατεία από τη δική μας πλευρά με αποτέλεσμα τελικά τέτοιου είδους προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις να διακοπούν. Από την άλλη όμως πλευρά νομίζω πως θα πρέπει να καταστήσουμε σαφέστατο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, εφαρμόσει κάποια στοιχεία της δήλωσης του Ιουλίου. Ε, ένας, ε, ε, ακούστηκε ένα αστείο από την πλευρά ενό εκπροσώπου τη Επιτροπή ότι από τον Ιούλιο η Επιτροπή μόνο σόγια Ε, νομίζω ότι τα όσα έχουμε κάνει από τη δική μας πλευρά μπορούν να δείξουν και στην, ε, προς τον πρόεδρο Τραμπ ότι πραγματικά εμείς έχουμε την, ε, την διάθεση να συνεργαστούμε. Πάντως ε, ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που ανέφερα μια σειρά από μια από συνάδελφοι είναι ότι, ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέψουμε στου Αμερικανού να διασπάσουν το κοινό μα μέτωπο ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακολουθώντα αυτή τη γραμμή, θα πρέπει ακριβώ να δώσουμε την κατάλληλη εντολή στην Επιτροπή, διατηρώντα την απαραίτητη διαφάνεια και διατηρώντα ένα κοινό μέτωπο, έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρανοήσει ευθύ εξ αρχή. Προκειμένου δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια μικρά βήματα και να μην συνεχιστεί ο κινησμό που εσεί κατά μα. Ευχαριστώ, λέω. ο πρόεδρο. Ζαν Λουκ, θέλει το λόγο για 10 λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρο θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα, δηλαδή ε, τον ε, Σύρο και τον χάλβα, Νομίζω πως από τον τελευταίο Ιούλιο αυτό που είπαμε ήταν ότι θέλουμε να ε, επιλύσουμε αυτό το ζήτημα, αλλά δεν υπήρξε καμία προσπάθεια από την Αμερικανική πλευρά να επιληθεί τον λόγο ζήτημα. Υπάρχει μια ισορροπία σε ό,τι αφορά τα αντίμετρα τα οποία εμεί ελάβαμε από τη δική μα πλευρά, ε, και τελικά ε, το αποτέλεσμα αυτών των μέτρων και αντιμέτρων ήταν πιο αρνητικό για την αμερικανική πλευρά γιατί ε, ο, η τιμή τους ε, χάλιβα αυξήθηκε περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σύγκριση με τους δεσμούς που είπαμε. Πάντως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα προτού ξεκινήσουν κανονικά οι διαπραγματεύσεις. Ε, σε ό,τι αφορά ε, την ε, απειλή που ακούσαμε, σε ό,τι αφορά την επιβολή δασμών, σε ό,τι αφορά τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, ας δούμε τι θα γίνει από, από εδώ και πλευρά. Η δική μας δήλωση είναι σαφής. ότι δηλαδή δεν μπορεί να περιλαμβάνεται κάτι το οποίο θα αντίκειται στο πνεύμα της συμφωνίας, εκτός και αν υπάρξει παραχώρηση από τη συμφωνία κάποιε από τι δύο πλευρέ. Δεν ξέρουμε δηλαδή αν θα υλοποιήσει αυτή την απειλή του ο πρόεδρο Τραμπ ή όχι. Αν το κάνει όμω, φυσικά αυτό θα σημάνει αυτόματη διακοπή των διαπραγματεύσεων. Θα πρέπει λοιπόν εμεί να δείξουμε αυτοπεποίθηση, να δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί και να θυμηθούμε ότι ήμασταν διατεθειμένοι να αντιδράσουμε απέναντι σε τέτοιου είδου μέτρα. Δηλαδή, είμαστε ω Ευρωπαϊκή Ένωση ε, εκείνοι οι οποίοι λάβαμε τα ισχυρότερα αντίμετρα άμεσα και σε ό,τι αφορά ε, το χάλιβα και σε ό,τι αφορά άλλα μέτρα. Οπότε έχουμε δείξει στους Αμερικανούς ότι είμαστε διατεθειμένοι να αντιδράσουμε. Και νομίζω πως αυτά τα αντίμετρα στο χάλιβα οδήγησαν στην επιτυχή έκβαση των συνομιλιών του Ιουλίου και την κοινή δήλωση. Ε, και ούτως ή άλλως δεν νομίζω πως ο πρόεδρος ε, Τραμπ ε, πριν από τα midterm elections περαιτέρω ήθελε περαιτέρω ε, συγκρούσεις. Πάντως σε ό,τι αφορά το να μπορέσουμε να έχουμε μία σε βάθος και διευρυμένη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να ε, συναυθεί μια τέτοια συμφωνία μια ε, χώρα η οποία δεν συμμετέχει ε, στη Συμφωνία των Παρισίων. Και θα συμφωνήσω με την κυρία Τιντάλινγκ σε αυτό που ανέφερε σχετικά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά αγαθά, του σχετικού δασμού, πράγματι αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο μια συμφωνία αυτή. Αλλά τελικά ε, ε, ε, σε τυπικό επίπεδο έχουμε πιο τομεακού χαρακτήρα επιμέρους συμφωνίας από ό,τι με αυτή. Ε, και αν εξαιρέσουμε τα αυτοκίνητα από αυτό το εμπόριο θα βρισκόμαστε στο 85% του συνόλου του, του διμερού εμπορίου. Δεν λέω ότι οπωσδήποτε θα υπάρξει αποκλεισμό των αυτοκινήτων, αλλά σε κάθε περίπτωση ένα κομμάτι τη αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή των, των σχετικών αγαθών, θα εξαιρεθεί από την ε, συμφωνία. Και υπάρχουν, για παράδειγμα, κάποια συγκεκριμένα ανταλλακτικά Ε, για τα ε, φορτηγά για παράδειγμα και φορτηγά στα οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα και στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τώρα το δευτεροβάθμιο όργανο προσφυγών, το Appellate Body, δεν απομένει πολύς χρόνος μέχρι τις ε, συζητήσεις στη Γενέβη να δούμε κατά πόσο θα είναι παραγωγικές εν λόγω συνομιλίες. Ε, ε, ε, αυτή τη στιγμή η Αμερικανική πλευρά έχει βέβαια αποδεχτεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ωστόσο, εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Πάντως, ε, ε, θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει εν λόγω συνομιλία, όπως στη Γενέβη, όπως έγινε και σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τι κρατησίε ενισχύσει Capital όπου δηλαδή είχαμε αρκετά καλές ε, ε, διαπραγματεύσεις πριν από δύο εβδομάδες ε, στην Ουάσιγκτον. Για το χρονοδιάγραμμα που ρωτήσατε, εφόσον υπάρχει συμφωνία και έχουμε εντολή διαπραγμάτευσης για τα δασμολογικά στα βιομηχανικά είδη, αυτό θα μπορούσαμε να το διαπραγματευτούμε πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ιδιαίτερα περίπλοκα δύσκολα ζητήματα και παρότι δεν έχει καμία σχέση είχε γίνει δουλειά υπό την TTIP και στις αξιολογήσεις συμμόρφωσης Και στα δοσμολογικά, όπω έλεγα προηγουμένω η βασική δυσκολία θα ήταν η αυτοκίνητο βιομηχανία. Για τους κανόνες προέλευσης ε, και σε κάποιε πτυχέ των κλωστοϊφαντουργικών επίση έχουμε επιμέρους ζητήματα, αλλά θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε τώρα για την ερώτηση που έγινε για τις ε, κυρώσεις, τις εξοεδαφικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ως Γενικός Διευθυντής Εμπορίου δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Η κυρία Μογκερίνη και η ομάδα της εργάζεται για να περιορίσει τον αρνητικό αντίκτυπο. Είχαμε κάποιες ε, επιτυχίες για την άρση συγκεκριμένων κυρώσεων όχι επειδή βέβαια συμπαθούμε τον κύριο Νταριπάσκα ή τον κύριο Πούτιν αλλά επειδή θα είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα για την βιομηχανία αλουμινίου και των προϊόντων αλουμινίου που χρησιμοποιούνται και στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε άλλους τομείς. Ήταν ένα δύσκολο θέμα στην Αμερικανική Βουλή, αλλά τελικώς δεν τον μπλοκάρισαν. Για το 232 δεν πρόκειται για νομοθετική πράξη, αλλά εκτελεστική εντολή της αρμόδιας διοίκησης και για τα γεωργικά το Κογκρέσο πιέζει αλλά πρόκειται για διέξοδο και για πολιτικούς λόγους πρώτον αλλά και ε, γιατί γνωρίζουμε ότι είναι πιο δύσκολο για μας από ό,τι για τους Αμερικανούς γιατί όπως είχαμε πει στο πλαίσιο της TTIP δεν μπορούν να κινηθούν καθόλου. Δεν είναι διατεθειμένοι να κινηθούν καθόλου. Επομένως επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση για τα φυτοϊγειονομικά. για τα γάματα φόμικρον ε, και συγκεκριμένες επεξεργασίες πουλερικών ε, εμείς ε, προασπιζόμαστε την αυτονομία τη ρυθμιστική μας και την προστασία βεβαίως των καταναλωτών και των πολιτών μας. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφισημία εδώ. Πάντως δεν πρόκειται, δεν δεχόμαστε να διαπραγματευτούμε όταν κάποιος κρατάει ένα πιστόλι στον κρόταφό μας. Γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και σε αντίμετρα. και σε κλιμάκωση. για την παρατήρηση που έγινε ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε μια ευρύτερη συμφωνία, μια πληρέστερη συμφωνία. Ε, ναι, αλλά αυτό θα προϋπέθεται κάποια ανταλλάγματα, το οποίο δεν έγινε στην TTIP. Και έχουμε και τη Συμφωνία των Παρισιών για, το, για την κλιματική αλλαγή και τις αποκλήσεις εκεί. Το βασικό όμως πρόβλημα και για τα γεωργικά και τα τρόφιμα είναι ότι αυτό που θα συνέβαινε είναι ότι θα στοχοποιούνταν συγκεκριμένα προϊόντα γεωργικά μας, το κρέας, τα πουλερικά, το χοιρινό. Διότι στοχεύουν σε πρώτες ύλες, σε βασικά αγαθά, οι Αμερικανοί, Υπάρχουν τα θέματα των NTB, των δεσμολογικών, αλλά επειδή εμείς κυρίως εξάγουμε υψηλής ποιότητας επεξεργασμένα προϊόντα, από αυτό προκύπτει το πρόβλημα. Δεν μπορούμε λοιπόν τον διάμεσο αυτό τομέα να τον καταστρέψουμε μέσω ε, πολύ αυξημένων εισαγωγών. Μπορούμε λοιπόν σε διάφορους τομείς να βρούμε κάποιες επιμέρους ε, συμβαστικές λύσεις, αλλά όχι εδώ. Δεν βλέπω κάποιο περιθώριο. Τώρα, για την κυρία Ντάλιν και την, ε, την εντύπωση που δίδεται είναι σημαντικό θέμα, αλλά δεν μας φοβίζει. Είχαμε τις κοινέ δηλώσεις που κάπως αποκλιμάκωσαν ε, την ατμόσφαιρα αλλά μένουμε στη θέση μας και καθότι στην ε, γραμμή που τηρούν οι Αμερικανοί δεν τηρούν τις κοινέ ε, αυτές δηλώσεις, πράγμα που εμείς κάνουμε, δεν μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε. Γιατί στον ε, κήπο των φίλων ο πρόεδρος Τραμπ διάβασε επιμέρους τμήματα των κοινών αυτών δηλώσεων, τα οποία δεν τηρεί. Το θέμα της προστασίας των δεδομένων δεν το συζητούμε ποτέ. Έχουμε και νέο μορφότυπο. και τις ε, διαδικασίες εντοπισμού που συνδέονται με τα δεδομένα αυτά. Δεν διαπραγματευόμαστε όμως καθόλου διμερώς για τα θέματα αυτά την Παρασκευή θα υπάρχει και μια συζήτηση e-commerce στον Τάβος και ελπίζουμε να έχουμε πολλούς συμμετέχοντες αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εμπίπτει στην διαπραγμάτευση αυτή. Δεν μιλούμε για TTIP, δεν μιλούμε για συζητήσεις ε, ε, του περιθερίου ή του διαδρόμου αλλά για ένα πλαίσιο που θα μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις και τους δύο, χωρίς να είναι τόσο ευρέω φάσματος. Άκουσα και κάποια καλά λόγια για την εμπιστοσύνη που δείχνεται στην Κομισιόν αυτό με ευχαριστεί, λέει ο μιλητής. Θα δούμε τώρα πότε θα έχουμε αυτή την διαπραγματευτική οδηγία. Ε, καλό θα ήταν να έχουμε το συντομότερο δυνατόν, ώστε να διαβιβάσουμε το μήνυμα ότι έχουμε πολιτική στήριξη για, την, ε, για το joint statement και ώστε να περιμένουμε τη δική τους κίνηση μετά από αυτό. Να σε ελπίσουμε ότι μια τέτοια διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης λόγω της αβεβαιότητας της δασμολογικής στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Φαντάζομαι ότι δεν μακρηγόρησα ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο επιπλέον παρατηρήσεις σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος. Έχουμε εκλογέ γρήγορα όπως ξέρετε και θα λείπουμε από τις Βρυξέλλες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και ίσως και Ιούλιο. Προβλέπετε να γίνονται διαπραγματεύσεις αυτό το τετράμινο. και το θέμα της ε, διάδοχης κατάστασης στην εντολή για το TTIP είναι υποσυζήτηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικές ε, εντολές. Καταρχάς δεν έχει ακυρωθεί η εντολή για το TTIP. Αλλά πριν το αναζωογονήσουμε για μια ακόμη φορά, κάτι το οποίο δεν γίνεται μάλλον σε αυτή τη φάση, δεν το συνιστώ τουλάχιστον, θα δούμε στο τέλος Ιουλίου αν θα είναι δυνατόν να δώσουν ορισμένες εξηγήσεις ε, για το πάγωμα αυτών των συζητήσεων. Το θέμα είναι λοιπόν πότε και εάν η Αμερικανική κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς ε, και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε μπορέσει να βρει κάποιες λύσεις αν θα μπορέσει να κάνει κάποια βήματα στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Δεν μιλάμε για το τοπικό περιεχόμενο, στην περίπτωση που υπάρχουν δημόσιοι διαγωνισμοί και προμήθειες που χρηματοδοτούνται από ομοσπονδιακά χρήματα και πιστώσεις γιατί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην βρίσκονται στο, εσω... ίδιο επίπεδο εν πάση με τις αμερικανικές επιχειρήσεις Το Jobs Act ε, έτσι και αλλιώς είναι πολύ πιο περίπλοκο, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, υπάρχουν ε, κάποια γενικότερα θέματα στα οποία θα μπορούσαμε να βρούμε μια κάποια λύση όπως οι μεταφορές. Από την άλλη υπάρχουν κάποιες εξειδικευμένες δραστηριότητες ε, πάνω στις οποίες δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να προβλέψουμε τις εξελίξεις. Ας πούμε η βυθοκόρηση, εκεί δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Τώρα, για τα γεωργικά προϊόντα οι διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Υπάρχουν συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους έχουμε σοβαρές διαφορές, όπως είναι η ζάχαρη. Σε επίπεδο νομικό, όπως είπαμε λοιπόν, η εντολή είναι ενισχύ. Από την άλλη δεν υπάρχει πολιτική ε, ε, όθηση ούτε για μένα είτε για τους διαδόχους μου για να μπορέσουν στην παρούσα φάση να κάνουν κάτι. Τώρα για τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Ιούλιο. Ας πάρουμε την οδηγία για τη διαπραγμάτευση από το Συμβούλιο. Ελπίζω να περιλαμβάνει και τις δικές σας συστάσεις. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν. και θα δούμε αν πράγματι υπάρχει προσπάθεια από κοινού και από τις δύο πλευρές Είναι σαφές ότι ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες επαφές ε, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, αλλά στον δαμολογικό τομέα οι διαφορές απόψεων είναι σαφές ότι είναι πολύ μεγάλες και δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Και έτσι κι αλλιώς οποιαδήποτε απόφαση και να ληφθεί είναι επίσης σαφές ότι το επόμενο κοινοβούλιο που θα σας διαδεχθεί θα πρέπει να επικυρώσει τις αποφάσεις. Ε, πάντως δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για τα επιμελητιακά κομμάτια αυτής της διαδικασίας. Καλώς θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή και θα συναντηθούμε εκ νέου. Λοιπόν, στην περίοδο που συζητάμε τα του Brexit, το να ολακληρώσουμε ε, τα θέματα των σχέσεων με την Ελβετία έχει αρκετό ενδιαφέρον και γι' αυτό θα δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μόλις ολοκληρώσαμε το πλαίσιο διαπραγματεύσεων με την Ελβετία, θεωρούμε ότι καλό θα ήταν να ενημερωθεί η Επιτροπή ΙΝΤΑ εγκαίρως. Η δική μου έκθεση ε, είχε ολοκληρωθεί πριν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά η συμφωνία επικαιροποιεί κάποια τμήματα ελευθέρων συναλλαγών από τη συμφωνία που είχαμε του 1992 και από κάποιες επιμέρους διμερείς συμφωνίες που είχαμε πιο πρόσφατες. Πολλοί από τους τομείς στους οποίους έχουμε συναλλαγές με την Ελβετία δεν του 1972... Ε, διορθώνει ο Διερμηνέας ε, γιατί αυτή η συμφωνία δεν συμπεριλάμβανε λοιπόν πάρα πολλούς τομείς τώρα πλέον έχουμε διευρύνει το πλαίσιο με νέους κανόνες για την τελωνιακή συνεργασία όπως και για την πνευματική ιδιοκτησία και τις δημόσιες προμήθειες. Καθότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις, θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο να μετατραπεί η έκθεση αυτή σε σύσταση, η γνωμοδότηση σε σύσταση, σχετικά με κάποιες από τις πτυχές που δεν συμπεριελήφθησαν τελικά στη συμφωνία. Για παράδειγμα, καλό θα ήταν να επανεξετάσουμε την γεωργική συμφωνία και να μην έχουμε εμπορικά εμπόδια, ιδιαίτερα για τους ελέγχους και τις αναγνωρίσεις γεωγραφικής προέλευσης. Τέλος, ε, θεωρώ ότι θα πρέπει ολοκληρωμένα να δούμε το θέμα των εργαζομένων ε, με δεσμευτικές διατάξεις για τις συνδίκες εργασίας και των μετακινούμενων εργαζομένων, ένθεν κακήθεν των συνόρων. γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα για πάρα πολλούς ε, ε, Ευρωπαίους πολίτες που βοηθούν στην οικονομία της Ελβετία. Οι τώρα. Γιατί την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Εγώ εργάζομαι στην υπηρεσία, στην ομάδα που ασχολείται με την Ελβετία στην ΙΕΔ που είναι πολύ σημαντικό σε διάφορους τομείς για το κλίμα, το περιβάλλον, ε, τα εκπαιδευτικά και την ελβετική συμμετοχή στην περιοχή Σέγγεν και στην εσωτερική αγορά. Ήδη ακούσαμε ότι η εμπορική σχέση αυτή είναι πολύ στενή. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις και χάρη στην Συμφωνία ε- Ελεύθερης Μετακίνησης έχουμε περί το 1,4 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που ζουν και εργάζονται στην Ελβετία και περί τους 450.000 Ελβετούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης έχουμε 300.000 περίπου εργαζομένους που μετακινούνται προς την Ελβετία για να εργαστούν καθημερινά. Μας συνδέει ένα ευρύ φάσμα διμερών συμφωνιών Ακούσαμε για την FTA του 1972, η οποία περιορίζεται σε εμπορικά και βιομηχανικά αγαθά. Υπάρχουν συμφωνίες συμμετοχής εσωτερικής αγοράς στις αερομεταφορές, αμοιβαία αναγνώριση, αξιολογής συμμόρφωσης, γεωργικά. Βέβαια έχουμε και κάποιους περιορισμούς και ελλείψεις που οφείλονται κυρίως στο γεγονός ε, της παλαιότητας ακριβώς του αρχικού πλαισίου συμφωνίας. Η FDA δεν καλύπτει τα γεωργικά αγαθά. Έχουμε επιμέρου συμφωνίες που δεν έχουν απελευθερωθεί με εξαίρεση το τυρί. το IPR, η εγκατάσταση, οι αναφορές στην κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση δεν συμπεριλαμβάνονται σε διάφορους από τους τομείς, δεν έχουν εξυγχρονιστεί δηλαδή αυτέ οι συμφωνίες και έχουμε και κάποιες περιοχές τις οποίες θεωρούμε ασύμετρη τη σχέση. Δεν έχουμε γενική συμφωνία για τις υπηρεσίες και μόνο περιορισμένη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Σε γενικότερο πεδίο, οι διατάξεις ε, ώστε να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο για τις κρατικές ενισχύσεις, για παράδειγμα, και την επίλυση διαφορών, είναι κάτι που μας λείπει. Έχουμε μόνο διπλωματικές επαφές για την επίλυση διαφορών μέχρι στιγμή. Όπως ακούσαμε από το 2014 είχαμε διαπραγματεύσει σε ε, μια συμφωνία θεσμικού πλαισίου για να πληρωθούν αυτά τα κενά, κάποια από αυτά τα κενά. Στις 23 Νοεμβρίου πέρυσι οι διαπραγματευτές ε, συμφώνησαν σε ένα τελικό κείμενο το οποίο υποβάλλεται προς διαβούλευση από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας. Αυτό θα είναι αμοιβαία υποφελές και θα δημιουργεί και μια ασφάλεια δικαίου για τους ε, φορείς και χρήστες της αγοράς. Θα έχουμε καλύτερη απορρόφηση του κεκτημένου σε διάφορες ε, περιοχές με, έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, διαφορών και προσφυγής στο δικαστήριο για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα έχουμε έναν ενισχυμένο λοιπόν μηχανισμό για, για να επιλύουμε διαφορές για κενά που είχαμε και που μας ενοχλούσαν για πολλά χρόνια στην εμπορική σχέση, την οικονομική σχέση με την Ελβετία. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας απέστειλε την πρόταση αυτή που, είχε, που είχαν συμφωνήσει οι διαπραγματευτικές ομάδες ε, προς διαβούλευση, αλλά δεν επικύρωσαν επισήμω τη συμφωνία αυτή. Επομένως, υπό τη δική μας οπτική γωνία είναι πολύ σημαντικό στο τέλος αυτής της περίοδου συζήτησης και διαφήνισης το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο να λάβει, να τοποθετηθεί επισήμως επιτέλους και να το υποβάλει στο Κοινοβούλιο προς επικύρωση. Και ένα σύντομο σχόλιο για το σημείο 7, για τα χαλιβουργικά. Οι βιομηχανίες μας είναι διασυνδεδεμένες, αλλά χρειαζόμαστε πολυμερή μέσα ή ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ που να μην είναι διακριτική μεταχείρισης. Επ' αυτού ίσως να χρειαστούν κάποιες περαιτέρω ανταλλαγές με τους Ελβετούς. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Now the Ευχαριστώ. Ισχυώδη συζητητέ ε, τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Βεγγίν και τον, την του και ε, επιχαίρουμε από την πλευρά τη δική μα ομάδα ότι φτάσαμε σε μια συμφωνία μετά από 1,5 χρόνο διαπραγματεύση και μετά από, την, ε, από μεγάλες προσπάθειες που έγιναν βέβαια και την ε, βούληση που υπήρξε σε πολιτική επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω πω θα επιτύχουμε περισσότερη ασφάλεια δικαίου για όλους. Και μην ξεχνούμε ότι το 52% ε, το 52% των εξαγωγών της Ελβετίας κατευθύνονται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 72% των εισαγωγών της ε, προέρχονται από αυτήν. Ε, από τότε λοιπόν που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις είχαμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε το κείμενο Αλλά είναι ε, παράξενο το γεγονό ότι δεν υπήρξε δημόσια διαθέσιμο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση το εν λόγω κείμενο και χρειάστηκε να το ζητήσουμε από την ελβατική κυβέρνηση. Ε, Εμεί ε, θα εξετάσουμε την, ε, το ενημερωμένο κείμενο τη Συμφωνία. Πάντως είναι σημαντικό το να τονίσουμε ότι το εν λόγω κείμενο, το οποίο δηλαδή συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο, είναι οριστικό και δεν θα ξανατεθεί προ διαπραγμάτευση. Νομίζω πω τέσσερα χρόνια διαπραγμάτευση ήταν υπεραρκετά. και αναμένω να ακούσω και του υπολείπου συναδέλφου προ το πώ θεωρούν και εκείνοι πως μπορεί να ε, εξυγχρονιστεί ε, περαιτέρω αυτή η συμφωνία. Ο κύριος Ντάτη τώρα από, το, από τους Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ε, αυτό το σχέδιο είναι με καλή βάση για εργασία και είναι πολύ σημαντικό γιατί θα συμπεριλάβει πέντε τομεακές συμφωνίες που διέπουν σήμερα την σχέση μας με την Ελβετία. Θα έχουμε λοιπόν μια πιο αποτελεσματική υλοποίηση των διατάξεων για την πρόσβαση στην αγορά των ελβετικών επιχειρήσεων. Και μιλούμε για ε, στρατηγικό συνεργάτη, δεύτερο για τις υπηρεσίες, σε περιοχή στην οποία έχουμε θετικό ε, ισολογισμό με τους Ελβετούς. Προσπαθούμε να έχουμε όσο υψηλότερο επίπεδο ολοκλήρωσης έχουμε προς το κεκτημένο Έχουμε τα, την εμπορία γεωργικών προϊόντων μαζί με την προστασία γεωγραφικών προελεύσεων όπως και για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών που είναι ένα από τα πιο δύσκολα και αντιφατικά ζητήματα σήμερα. Και έχουμε και μία φάση συζήτησης για μελλοντικές συμφωνίες και ενεργειακές. Η συμφωνία λοιπόν έχει τη δυνατότητα να επιφέρει νέες καινοτομίες και στο εμπορικό επίπεδο που και τα δύο μέρη συμφώνησαν ε, να δεσμευτούν όπως και για τον εξυγχρονισμό των συμφωνιών για τις δημόσιες προμήθειες του 2020 που σήμερα έχει δυνατότητα να προχωρήσει και πέραν των διατάξεων του ΠΟΕ και τη FTA του 72 που δεν προλέπει ε, μηχανισμό επίλυση διαφορών. Εμείς ε, θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίε για κάποιες ε, θεματικές που θεωρούμε ότι σημαντικό να αναφερθούν. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο και ελπίζω και είμαι βέβαιο ότι μπορούμε να συνεργαστούμε καλά σε αυτό το φάκελο. Ο κύριο ε, Σταμπάτη τώρα για το ECR. Κύριε Πρόεδρε, ε, εξέτασα αυτή την ε, θεσμική συμφωνία πλαίσιο και θεωρώ πως σε μια μεγάλη πολιτική δύναμη επιβάλλει στον ε, πιο αδύναμο, αν θέλετε, ε, εταίρο της, ε, τους δικούς της όρους. Για παράδειγμα, το ζήτημα της ερμηνείας της νομοθεσίας από την πλευρά του δικαστήριου, του Ευρωπαϊκού ε, να σας πω ότι έχω κάποια εμπειρία σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ευρώ και θα πρέπει να πω ότι το δικαστήριο ε, ουσιαστικά τι κάνει. Ε, κάνει ακολουθεί μια λογική ανάποδη. Δηλαδή, ε, καταρχήν ορίζει το τι θέλει να επιτύχει και στη συνέχεια προσπαθεί να δικαιολογήσει την απόφαση του με βάση αυτό που θέλει να επιτύχει. Από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, σε ό,τι αφορά την αρχή τη επικορικότητα. τι λέει η αρχή της επικορικότητας Ότι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη μπορούν να, να αποφασίζουν πλέον δεδειγμένοι ε, για τη λύση που χρειάζεται ο πολίτη. Αυτή είναι η βασική αρχή της ε, επικουρικότητας. Άρα λοιπόν όταν λέμε ότι θα πρέπει να ακολουθούμε πάντοτε την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα συστήματα διαφωνών, τότε ε, ουσιαστικά παραβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας. Ε, σε ό,τι αφορά τα συστήματα τώρα ε, ε των πληρωμών συνοχής. οι πληρωμές συνοχή δεν υπήρχαν πριν από κάποια χρόνια. Αυτό είναι αναπτυξιακή ε, βοήθεια, αναπτυξιακή ε, πολιτική. Όταν είχαν ε, προσχωρήσει κάποια κράτη-μέλη προηγουμένω, αυτό είχαμε πει όταν λέγαμε για παράδειγμα ότι δεν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξη. Και από εκεί και μετά. σε ό,τι αφορά την ισοδυναμία, σε ό,τι αφορά τις χρηματογορές σε περίπτωση που δεν υπάρξει μία σύναψη αυτής της συμφωνίας ε, νομίζω πως ε, είναι λίγο υπερβολικό αυτό το οποίο αξιώνουμε. Δηλαδή, εάν αυτή η συμφωνία πλαίσιο τεθεί ε, πρόσφυση σε δημοψήφισμα από τους πολίτες δεν θα συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ψηφών των πολιτών γιατί αυτό που θα αναφερθεί είναι υπάρχει ένας ισχυρότερος εταίρος ο οποίος επιβάλλει τη βούλησή του σε ένα πιο αδύναμο σε ένα λιγότερο ισχυρό εταίρο οπότε νομίζω πως θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτό το κείμενο της συμφωνίας έτσι ώστε να καταστεί αποδεκτό από την πλευρά της Ελβετίας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για τους πράσινους ο ε, Καρμπούχνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, σκέψεις που ακούστηκαν τώρα, εμφιβολίες δηλαδή και δυσπιστία και το γεγονός ότι ενδεχομένως να επιβάλλουμε τη δική μας ευούληση στην Ελβετία, Εντάξει, ε, ε, δεν μπορώ να υπερασπιστώ αυτή τη θέση. Πάντως, ε, ό,τι αφορά τη διαδικασία, να πω ότι άκουσα ότι στις 7 Δεκεμβρίου καταλήξαμε σε μια συμφωνία στην οποία δηλαδή κατέληξε ως διαπραγματευτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την οποία μας λέει ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω. Μα αν έτσι έχουν τα πράγματα, δεν ξέρω αν έχουν έτσι, αλλά αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε τι χρειάζεται η περαιτέρω συζήτηση που κάνουμε αφού δεν μπορεί να αλλάξει το κείμενο. Και πού βρίσκεται αυτό το κείμενο. Δεν το έχω λάβει εγώ από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πρέπει να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είχε επαναληφθεί στο παρελθόν. Πρόκειται δηλαδή για ε, πλήρη υποτίμηση και περιφρόνηση ε, της, ε, του δημοκρατικού ελέγχου από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατά συνέπεια δεν μπορώ να είμαι θετικά απέναντι σε μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ πρόεδρο. Πράγματι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τη Γενική Διευθύνση Εμπορίου και έχουμε συνέψει μια συμφωνία σε ό,τι αφορά την ε, ε κοινή πρόσβαση στις πληροφορίε και στα έγγραφα. Αλλά εδώ δεν ακολουθήθηκε αυτή η συνήθιση ε, γραμμή που ακολουθεί η Γενική Διεύθυνση και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, και η δική μου τιμή ή και ευθύνη ή οτιδήποτε άλλο είναι εδώ και δύο χρόνια να διαπραγματεύομαι με το Συμβούλιο, με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προκειμένου ε, αυτή η συμφωνία που έχουμε συνάψει με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να αποτελέσει το υπόδειγμα για τη σχέση μα με όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Με το Συμβούλιο δηλαδή, με την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ωστόσο και οι δύο αυτοί εταίροι έχουν επιφυλάξει σε σχέση με αυτή τη συμφωνία και δυστυχώ αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Αλλά ίσω η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση μπορεί να δώσει κάποιε απαντήσει στα σχόλια αυτά που ακούσαμε από του συναδέλφου. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Uh, uh, Φαίνεται λίγο ασυνήθιστο, αλλά η διαπραγμάτευση αυτή έτσι κι αλλιώ ήταν ασυνήθιστη από την αρχή μέχρι το τέλος. Πάντως καταλήξαμε κάπου με τον Ελβετό διαπραγματευτή μετά από τις 23 Νοεμβρίου. Θεωρήσαμε ότι είχε κλείσει, για μας έχει κλείσει. Ο Ελβετό Διαπραγματευσής ζήτησε την έγκριση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Συνομοσπονδία. και ε, καταλάβαμε ότι σε εκείνη τη φάση δεν θα υποστήριζαν τη συμφωνία αυτή αλλά θα ξεκινούσαν μια δημοψηφισματική διαδικασία. Πρόκειται για μια ειδικού τύπου διαδικασία μάλλον η οποία ε, καλύπτει την αναζήτηση της γνώμης εμπορικών εταίρων, οικονομικών εταίρων, κοινοβουλίων, τοπικών αρχών. Θα κρατήσει η διαβούλευση αυτή ένα τρίμηνο και μετά θα πάρει απόφαση το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. για να υποστηρίξει ελπίζουμε τη συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει με τους Ελβετούς διαπραγματευτές. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση νομικά θα έλεγα λίγο σε κρεμότητα και γι' αυτό ακριβώς δεν είχατε και επίσημα το αντίγραφο της τελικής συμφωνίας. Αλλά είμαι στη διάθεσή σας γι' αυτό. <clears throat> Τιτσιάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους σκιώδεις συναδέλφους, εισηγητές, με τους οποίους ε, από κοινού εκφράσαμε τη δυσφορία μας για τις τελευταίες εξελίξεις. Κατανοώ εν μέρη αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έτσι και αλλιώς θα μπορούσε να διανεμηθεί η συμφωνία αυτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια τελική έγκριση από πλευράς της Ελβετίας. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω με τα σημεία που έθεσαν οι συνάδελφοι και θα προσπαθήσω να τα συμπεριλάβω στην τελική σύσταση. Καλώς. Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι 25 Ιανουαρίου, 6η απογευματινή. Παρακαλώ στα αγγλικά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί επί της ουσίας αρμόδια η ΑΦΕΤ ε, θα πρέπει να ψηφίσει στο τέλος Φεβρουαρίου και θα πρέπει να είναι έτοιμη μέχρι τότε η δική μας εμπασπεριτώση γνωμοδότηση. Λοιπόν, 25 Ιανουαρίου στα αγγλικά παρακαλώ. Οι σκιώδεις θα πρέπει να τα συζητήσουν αυτά αρκετά σύντομα. και ελπίζω 1η Φεβρουαρίου να ψηφίσουμε. Επίσης ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη η Επιτροπή τις ανησυχίες μας σε σχέση με την σωστή διαφάνεια και την σωστή ενημέρωση. Κλείνουμε το 6. Περνάμε στα 7 και 8. συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ. Χάουταλα, η συγγήτριά μας. 5 με 6 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εμένα μου είχαν πει το αντίθετο ότι είχαμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτική. Όπως είχαμε πει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, ε, εκλήθη να κάνω μια ιδιωτική ανοιχνευτική επίσκεψη στο Βιετνάμ. Πήγα τώρα στις αρχές Ιανουαρίου, ήταν χρήσιμη η συνάντηση και ήταν χρήσιμο θα έλεγα και για τις αρχές του Βιετνάμ να δουν ότι εμείς εκτιμούμε ιδιαίτερος αυτό το εμπορικό μέσο το οποίο προωθεί με σημαντικό τρόπο την αηφορία στην ανάπτυξη. Τελικά, οι συμφωνίες αυτές εθελοντικού τύπου συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της αποψήλωσης των δαθών συνολικότερα και η διαδικασία που οδηγεί στις αποφάσεις αυτές είναι μια διαδικασία διαπραγματευτική ιδιαίτερα σημαντική γιατί η κοινωνία των πολιτών παρακολουθεί τη διαδικασία και χαίρομαι να πω ότι στην περίπτωση του Βιετνάμ η διαδικασία αυτή <clears throat> σημείωσε ένα χωρίς προηγούμενο επίπεδο συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών κάτι το οποίο συνεισφέρει νομίζω σε πολλές αλλαγές στη χώρα και μάλιστα αλλαγές συστημικού τύπου. Η συνεργασία που είχαμε λοιπόν μαζί τους είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει και σε άλλες περιπτώσεις διαπραγμάτευσης που έχουν σαν στόχο τα δασικά προϊόντα. Είναι η πρώτη συμφωνία την οποία επεξεργαζόμεθα με μια χώρα η οποία ε, επεξεργάζεται ε, και η ίδια τα προϊόντα ξυλίας δεν είναι απλά παραγωγός δηλαδή. Οπότε ε, θα επανεξετάσει έτσι και αλλιώς την βιομηχανική της αυτή δραστηριότητα η Δημοκρατία του Βιετνάμ. Δραστηριότητα η οποία θυμίζω ότι είναι η τέταρτη σε επίπεδο ποσοτικό ε, στον κόσμο. Η επεξεργασία προϊόντων ξυλίας λοιπόν έχει πάρα πολύ ε, μεγάλες προοπτικές και συνεισφέρει ιδιαίτερο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Ήταν πάρα πολύ θετικό που το Βιετνάμ θέλει να διευρύνει τη δραστηριότητα αυτή αλλά με έναν αηφόρο τρόπο, έναν βιώσιμο τρόπο. Η εφαρμογή λοιπόν του VPA θα είναι μια σειρά θα έλεγα ενεργειών δύσκολων, μακρόχρονων ε, και θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι κάτι τέτοιο με την Ινδονησία χρειάστηκε 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Αλλά βλέποντας την αφοσίωση στην προσπάθεια την οποία επιδεικνύουν οι Βιετναμέζοι δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο. Ε, πρόσφατα το Βιετνάμ ήταν στο κέντρο μιας απαράδεκτης εμπορικής παράνομης δραστηριότητας προϊόντων ξυλίας ε, και τοπικά και σε σχέση ε, με ε, την Καμπότζη. Εμείς λοιπόν παρακολουθήσαμε την κατάσταση και είδαμε ότι ισχυρίζονται οι Βιετναμέζοι ότι είναι αποφασισμένοι να καταπολεμήσουν τις παράνομες αυτές δραστηριότητες και τη λαθρεμπορία προϊόντων ξυλίας ιδιαίτερα με προέλευση την Καμπότζη. Έχουν ε, επίσης ε, συμφωνήσει σε ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου ε, που απαγορεύει πλήρως την εισαγωγή παρανόμως υλοτομηθέντων προϊόντων και το Βιετνάμ θα είναι η πρώτη χώρα στην περιοχή και η τέταρτη χώρα στον κόσμο μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένε Πολιτείες και την Αυστραλία που θα αναλάβει αυτού του τύπου τις υποχρεώσεις. Πόσο μάλλον που το Βιετνάμα θέλει να εμπλέξει την κοινωνία των πολιτών στην παρακολούθηση των διαδικασιών αυτών και ένα από τα θέματα, που είναι ένα από τα θέματα στα οποία επιμένουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω τη σημαντική ε, δραστηριότητα της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ανόη. Υπό το φως λοιπόν και της τελευταίας αυτής αποστολής, εγώ σαν εισηγήτρια ε, θα συμπληρώσω ε, με επιπλέον συστάσεις την πρόταση εκθέσεως. Θα δείτε γραπτά τις εκθέσεις αυτές ταχύτατα έτσι ώστε το Βιετνάμ να χρησιμοποιήσει σωστά και ανοιχτά κριτήρια για τα προγράμματα αναγνώρισης. Να πω ότι επίσης και οι ενώσεις ε, βιομηχανικών ξυλίας, η ΧΑΟΑ, η οποία και αυτή, ε, η ένωση μάλλον αυτή, ε, συμμετέχει πλήρως στη διαδικασία. Θα υπάρξει επίσης και η απαιτούμενη συνεργασία ανάμεσα στο κεντρικό επίπεδο εξουσίας και τις περιφερειακές αρχές και θα στηρίξουμε εμείς από πλευράς μας τη διαδικασία αυτή. Η πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει στα πλαίσια των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας η συμφωνία αυτή να τύχει ε, ε, υψηλής ιεράρχησης από πλευράς μας και καταλήγω, χωρίς να ξεπεράσω πολύ τα 6 λεπτά, λέγοντας ότι είδαμε αρκετά θετικέ εξελίξεις στο Βιετνάμ. Η νέα νομοθεσία για την υλοτομία ε, ε, τέθηκε ισχύ στην αρχή του χρόνου ε, παγορεύει πλήρως την εισαγωγή όπως είπαμε παράνομης ξυλίας και θα πρέπει να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατόν να εφαρμοστεί ε, η συγκεκριμένη αυτή πρόβλεψη από τις αρχές του Βιετνάμ. Επισκεφθήκαμε την πρωτεύουσα της Καμπότζης σύντομα την Πνομπέ και ήρθαμε σε επαφή και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολίτων και είδαμε ότι το λόμπι της παράνομης ξυλίας έχει αρχίσει και δραστηριοποιείται εκ νέου αν και σε μικρότερη κλίμακα η Καμπότζη απαγορεύει δια νόμου εξαγωγές ε, προϊόντων ξυλίας. Έτσι κι αλλιώ οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή συνεπώ σε αυτό το επίπεδο είναι παράνομη και γι' αυτό δεν βλέπω γιατί το Βιετνάμ να μην θέσει σε ισχύ ένα μορατόριο ε, για την απαγόρευση της ε, εμπορίας ξυλίας ε, περιμένοντας το τίλα στην πλήρη συμφωνία συνολικά για τα προϊόντα ξυλίας ε, που θα τεθεί σύντομα σε ισχύ. Είχαμε λοιπόν καλές επαφές ε, και με το Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου και είμαστε βέβαιοι ότι το Βιετνάμ αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Ε, χαίρομαι εδώ γιατί ο κύριος Ζαχραντήλ ε, θα οργανώσει μια συνάντηση για το VPA ε, στα πλαίσια της επόμενης συνάντησης για το Βιετνάμ στις 4 Φεβρουαρίου και θα συμμετέχει και ο πρέσβης μας στο Χανόι και επίσης θα συμμετέχει και μία ΜΚΟ η οποία ελέγχει τα θέματα περιβάλλοντος στη συγκεκριμένη χώρα. Ελπίζω να οδηγηθούμε λοιπόν στην σύντομη επικύρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Η Σκιώδης τώρα. Ο κύριος Σάντι θα έχει λίγο πρόσθετο χρόνο διότι, έχει, διότι είναι Σκιώδης και για την ε, γνωμοδότηση για την ε, ανάπτυξη. Ο κύριος Προύστ ε, όμως πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Χάουταλα για την ποιότητα ε, του κειμένου της μελέτης της που περιλαμβάνει όλες τις στοιχές ε, που μας ενδιαφέρουν σχετικά με μια ρυθμισμένη, πλαισιωμένη σχέση για τα προϊόντα ξυλίας και την νόμιμη υλοτόμηση. θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε εδώ <clears throat> και τις ε, εμπορικές μας σχέσεις, αλλά να βελτιώσουμε και τις πρακτικές μας μέσω μιας ε, συμφωνίας που δεν είναι ακριβώς συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, <clears throat> και μερικές φορές ε, αναλαμβάνουν, προχωρούμε μάλλον στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών για λόγους κάθε άλλο παρά εμπορικούς. Αυτή εδώ η εθελοντική συμφωνία μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την όλη διαδικασία της παραγωγής και της λιωτόμησης ε, προϊόντων ξυλίας και εκφράζω την ικανοποίησή μου για, τις, ε, την καλή συνεργασία με τις Βιετναμέζικες Αρχές και συγχαίρω την εισηγήτρια για μια πολύ καλή έκθεση επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ. οι σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Γιώχιμ Σούστα. Η κυρία Μαρία Ρένα, η σκιώδης εισηγήτρια μας, ε, μου ζήτησε να διαβάσω ε, εκ μέρους της ε, μια σύντομη τοποθέτηση από πλευρά μας. Στα αγγλικά. Ευχαριστούμε λοιπόν για την μελέτη αυτή που είναι πολύ καλή βάση για εργασία. Νομίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει στο Βιετνάμ να αντιμετωπίσει πραγματικά την παράνομη εμπορία προϊόντων ξυλίας. Γνωρίζουμε το φαινόμενο αυτό και στην Καμπότζη και στο Λάος, αλλά και σε άλλες ε, χώρες που εξάγουν προς το Βιετνάμ. Ε, το Κονγκό είναι η τελευταία περίπτωση παράνομων προϊόντων ξυλίας, ε, δηλαδή εξαγωγής προς το Βιετνάμ. Επομένως η συμφωνία αυτή θα μας επιτρέψει απόλυτη διαφάνεια σε όλη την το πεδίο υλοποίηση και επιτήρησης. Και είναι πολύ σημαντική και για την κοινωνία των πολιτικών και τι τοπικέ κοινωνίε Θα μας επιτρέψει μηχανισμούς ε, που θα εξασφαλίσουμε καλύτερη υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου του Βιετνάμ. Μας φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το παράνομο αυτό εμπόριο σε όλη την αλυσίδα προμήθεια, επεξεργασία και πώληση εμπορία και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα την περιφερειακή διάσταση του προβλήματος. Εάν το Βιετνάμ προχωρήσει σε ισχυρή νομοθεσία, δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι γειτονικέ του χώρες έχουν σημαντικά φαινόμενα και παράνομης υλοτομίας και παράνομης επεξεργασίας. Εξού και οι τροπολογίε που θα υποβάλουμε, αλλά προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή συνεργασία με όλου του συναδέλφου σε αυτόν τον σημαντικό φάκελο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος ε, Σάραντι έχει έξι λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχουμε τρει φακέλους επί του Βιετνάμ στην προετοιμασία που δεν συνδέονται νομοθετικά ή διαδικαστικά αλλά επί της ουσίας γιατί εφόσον επικυρωθεί η FTA θα απελευθερώσει τα προϊόντα υλοτομίας και εξηλίας και είναι απαραίτητο να εξετάσουμε, να έχουμε ολοκληρώσει με το φάκελο αυτό προηγουμένως. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξή τρία. Καταρχάς τα όσα κάνει η κυβέρνηση του Βιετνάμ και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι είχαμε απτές εξελίξεις και βελτιώσεις μετά από μια αρκετά μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων που είχε ήδη ξεκινάσει το 2010 αν ακούσαμε καλά με διευκρινήσεις για το νομοθετικό πεδίο, για τις δασικές εκτάσεις και μια σημαντική διάταξη που ε, τέθη ενισχύ από 1η Ιανουαρίου και που απαγορεύει εισαγωγές από το Βιετνάμ παράνομων προϊόντων ξυλίας. Συμφωνώ ότι η επιβολή, η υλοποίηση των διατάξεων αυτών θα είναι το πιο σημαντικό θέμα. Για το επιχειρηματικό περιβάλλον στο Βιετνάμ και το πώς αντιδρούν οι επιχειρήσεις, και κατά πόσον θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο πλαίσιο, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε στενά κατά πόσον οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να εισαγάγουν εθελοντικά μέτρα συμμόρφωσης προς διατάξη αυτές και μόνο τότε θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα το τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι οι παράνομες εισαγωγές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν παράνομες εισαγωγές από Καμπότζη και Λάος κυρίως, αλλά όχι μόνο. Και από πιο μακριά έχουμε παράνομες εισαγωγές από την Αφρική. Από χώρες με υψηλό δίκτυ διαφθοράς και Πολεμικέ συγκρούσεις κάποιε φορέ. Επομένως θα πρέπει να εστιαστούμε στα μέτρα που θα αποτρέπουν την παράνομη εμπορική ροή προϊόντων ξυλία και από την Αφρική προς το Βιετνάμ. Ε, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να είναι αυτόματο και να γίνει άμεσα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. και με ικανοποίηση βλέπω και σημειώνω και την συμφωνία της συζητήτριας και σύντομα νομίζω ότι θα έχουμε έκθεση και από την ΔΕΒΕ που ήδη ε, επικύρωσε, ψήφισε χθε για την δική μου έκθεση. Σας ευχαριστώ κυρία Ρίς ε, για τους φιλελεύθερους. Ε, και η κυρία Λαλόντ, όπως και η προηγούμενη η Σκιώδης, θα ήθελε να ευχαριστήσει την κυρία Χάουταλα για το σχέδιο έκθεσης που είναι πληρέστε το θεωρούμε. Ε, περιγράφει πολύ καλά τις μεγαλύτερες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την υλοποίηση την ε, νομοθετική και την ε, επιβολή που θα πρέπει να έχουμε ώστε να έχουμε μια βιώσιμη συνεργασία στα προϊόντα ξυλίας παρακολουθώντας τις ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, για το Βιετνάμ, ε, πρέπει να προσέξουμε την δυνατότητα των βιετναμέζικων αρχών να σεβαστούν τον στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΠΑ και το θεματολόγιο 2030 τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Βιετνάμ για την υλοποίηση της συμφωνίας αυτής ε, αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια συνολική πλήρη συμμόρφωση προς τις ε, αξίες ε, της υπευθυνότητα που προσυπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ουσιώδου σημασία η σωστή υλοποίηση των διατάξεων αυτών για την πρόσβαση στην αγορά. Και υποβάλλουμε κάποιε τροπολογίε που πηγαίνουν προς το πνεύμα τη συγκήτρια, ώστε να έχουμε και τη συνεργασία των συνυπογραφών τη συμφωνία αυτή πέραν του Βιετνάμ και να έχουμε ε, ε, μια προσοχή στην ευρύτερη ε, περιοχή. Η Κίνα ιδιαίτερα πλήττεται από την παρανομία μπορεί ξυλίας, όπως θα πρέπει να γνωρίζουμε και η συμμετοχή μιας τόσο σημαντικής χώρας όσο η Κίνα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα ήταν μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Η σημαντική υλοποίηση της συμφωνίας κατά την κυρία Λαλόν θα πρέπει να περάσουν από απτές πράξεις σε όλη την αλυσίδα προμήθειας και εμπορίας τους, ε, τις υπεργολαβίες τρίτων χωρών ε, υποτένει αυτή η κυρία Λαλόντ υποστηρίζει το σχεδίο αυτό ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ λέω Πρόεδρος και τώρα για την ΚΟΕ. Yes, thank you, Mr. Chair. I speak on behalf of... Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ε, παίρνω το λόγο μέρο τη ε, Λόλα Σάντσε, η οποία δεν μπορούσε να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Η ομάδα μα, λοιπόν, υποστηρίζει τι δράσει ΕΦΛΕΚΤ, e αλλά το σχέδιο δράση, ειδικότερα στο πλαίσιο τη συμφωνία με το Βιετνάμ, θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα καταπολέμηση διαφθορά στον τομέα τη διασωκομεία, αν θέλουμε να είναι αποφασισματική αυτή η συμφωνία. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν υψηλότερη διαφάνεια, περισσότερη συμμετοχή, ανάληψη ευθύνη και καλύτερη εφαρμογή τη νομοθεσία στο πλαίσιο του ΦΛΕΚΤ ειδικότερα σε ό,τι αφορά την καλύτερη εφαρμογή της ε, ε, κοινοποίηση των πληροφοριών και μάλιστα πληροφοριών ε, που διατίθενται με τέτοιο τρόπο και με τέτοια γλώσσα που είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. Επίσης υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά τον ε, χώρο της κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο της FLECT. Ε, ε, θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν πάντοτε ανεξάρτητοι παρατηρητέ σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση της νομοθεσίας FLECT. Επίσης θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες δυνατότητες και στην δικαστική εξουσία για την άσκηση της δικής της, ε, ε, των αρμοδιοτήτων της. Επίσης ε, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι όλα τα VPAs, όλες οι σχετικές συμφωνίες περιλαμβάνουν μέτρα καταπολέμηση διαφθορά σε περίπτωση συγκρούσεων, έτσι ώστε οι διάφοροι παραγωγοί, αγροτικοί παραγωγοί, να μην υποβάλλονται σε αρνητικέ συνέπειε. Επίση, θα πρέπει να ασκηθούν πιέσει ώστε να υπάρξουν μεταρρυθμίσει στο ε, τομέα τη διακυβέρνηση, προκειμένου να τα καταπολεμηθεί η διαφθορά. Για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων, σε ό,τι αφορά τι χορηγίε. Θα πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν ε, ζητήματα διαφθοράς και ζητήματα διαφθάνειας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο σενό πλαίσιο του FLECT. Τέτοιου είδους μέτρα θα μπορούσαν να ε, περιλάβουν για παράδειγμα τον καλύτερο συντονισμό αυτών των χωρών FLECT ε, και των χωρών που δίνουν την βοήθεια όπως επίσης και συντονισμός αυτού του τομέα της πολιτικής με άλλες πολιτικές ειδικότερα στο πλαίσιο της καταπολέμησης του εξελίγματος βρώμικου ε, και επίσης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης τέτοιων ε, συμφωνιών με τρίτες χώρες θα πρέπει να ε, μειώνονται εδώ οι πιθανότητες σύγκρουσης συμφερόντων και θα πρέπει να εξασφαλίσετε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και η κατάλληλη πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ και ο λόγος τώρα στον κύριο Σαχαντήλ ως τον ε, αρμόδιο ε, από την πλευρά της Επιτροπής ΔΕΒΕ για το ίδιο ζήτημα των δηλαδή της σχετικής νομοδότησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, θα ήθελα να σας πω ότι με 17 τροπολογίες στο σύνολό τους εγκρίθηκε ομόφωνα χθες στην Επιτροπή ΔΕΒΕ η δική μου γνωμοδότηση. δύο εξαιρέσεις υπήρξαν μόνο σε ό,τι αφορά αυτές τις τροπολογίες, ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, μία τροπολογία σε ό,τι αφορά αυτές τις μάρτυρες του δημοσίου συμφέροντος ε, και την άλλη σε ό,τι αφορά το, την εφαρμογή, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα διαφάνειας. Αυτές οι δύο τροπολογίες δηλαδή δεν με έβρισκαν σύμφωνο, αλλά κατάφεραν να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ευχαριστώ. Ο κύριος Ούγκο Μαρία Σάλι. Ο επικεφαλής δηλαδή της μονάδας για τον Global Sustainability από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πάρει τώρα το λόγο για 5-6 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε ε, και εξότιμα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που υπόθηκε ήδη και από άλλους, δηλαδή υποστηρίζουμε τον συγκεκριτή και την υποστήριξη που εκφράζει απέναντι σε αυτή τη διαδικασία και ε, για το ενδιαφέρον που έδειξε, δηλαδή να μεταβεί στο Βιετνάμ ούτως ώστε να διαπιστώσει πώς έχουν τα πράγματα επί Με αυτόν τον τρόπο ενισχύσαμε και περαιτέρω τα μηνύματα τα οποία δώσαμε στο Βιετνάμ στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Ε, αναγνωρίζουμε όλες τις προκλήσεις ε, που αναφέρει ο ε, και οι σκιώδεις συγκητές, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τα μέτρα ελέγχου των εισαγωγών και επαλήθευση της στήριξη όλων των διατάξεων της ΦΔΕ και πλήρη συμμετοχή όλων stakeholders στο πλαίσιο της υλοποίησης και της παρακολούθηση της υλοποίησης της συμφωνίας. Προφανώς η δική μας δέσμευση που αναλαμβάνουμε είναι να συνεργαστούμε στενά με το Βιετνάμ στο πλαίσιο της ε, περίοδου υλοποίησης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι πράγματι αποκρίνεται το Βιετνάμ στις υποχρεώσεις του. Είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι το σχέδιο του ψηφίσματος ε, υπογραμμίζει αυτά τα στοιχεία ε, εμφατικά και αναφέρει μεταξύ άλλων για παράδειγμα ε, την ανάγκη για ανάπτυξη περαιτέρω νομοθεσίας, ε, νομοθεσίας η οποία θα αφορά σε ό,τι αφορά και την διασφάλιση της διαφάνειας και καταπλέμησης διαφθοράς και επίσης επιχαίρουμε το γεγονός ότι θίγεται εδώ το ζήτημα των εισαγωγών από γειτονικέ χώρε, αλλά όχι μόνο και από την Αφρική για παράδειγμα, γιατί η Αφρική αποτελεί μια σημαντική χώρα εισαγωγών ξυλία προ το Βιετνάμ. Θα συνεχίσουμε και σε αυτό το επίπεδο να παρακολουθούν από κοντά τα πράγματα. Είναι σημαντικό ε, το γεγονό ότι το Βιετνάμ ε, πρόσφατα υιοθέτησε ένα ε, σχέδιο εφαρμογής της Συμφωνίας ΕΒΠΕ στο 2021 και με αυτόν τον τρόπο ε, διασφαλίζει βέβαια και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά κονδύλια για την υλοποίηση της συμφωνίας ΕΒΠ. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται και η κατάλληλη παρακολούθηση από την πλευρά των stakeholders. Ε, ε, με αυτόν τον τρόπο βέβαια ανταποκρινόμαστε και στις ανησυχίες που εξφράστηκαν από την πλευρά διαφόρων ομιλητών σήμερα και σίγουρα θέλουμε να ε, κινηθεί το Βιετνάμ ε, το ταχύτερο δυνατό προς την ελοπίση ε, του συστήματος αδειοδότησης γιατί πράγματι θα βελτιώσει πολύ τα πράγματα αλλά με βάση την εμπειρία που είχαμε μέχρι τώρα είμαστε επιφυλακτικοί δεν ξέρουμε δηλαδή κατά πόσο το Βιετνάμ θα τηρήσει το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την θετική στάση που ακολουθεί η δική σας Επιτροπή αλλά και η Επιτροπή ΝΤΕΒΕ σε ό,τι αφορά αυτήν την ε, συμφωνία και αναμένουμε ε, την ταχεία ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Να επανέλθω λίγο στην, στο ιστορικό αυτής της υπόθεσης καλύπτουμε το σύνολο της παραγωγής και της παραγωγικής διαδικασίας, κυρίως για τα προϊόντα που προορίζονται προς εξαγωγή. Και προφανές είναι ότι για το Βιετνάμ η εξαγωγή ξυλίας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ποια είναι η αίσθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλύπτεται το σύνολο της παραγωγής. Καλύπτεται δηλαδή και η παραγωγή με, για προς εσωτερική κατανάλωση. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση του μηχανισμού παρακολούθησης. Το πρόγραμμα δράσης ΦΛΑΚ είναι κάτι το οποίο είχε σαν στόχο την βελτίωση της ε, διαχείρισης και της νομοθετικής δραστηριότητας του συνόλου του δασικού τομέα. καλύπτει στην ουσία δηλαδή την βιομηχανία ξυλίας, την υλοτομία και μιας και αυτού του τύπου οι εθελοντικές συμφωνίες είναι κατά βάση εμπορικές συμφωνίες, εξαρτάται από τη συγκεκριμένη χώρα αν θέλει να υποβάλει το σύνολο της δραστηριότητας στις απαιτήσει αυτές. Γενικά, οι χώρες εταίροι οι οποίοι έχουν συνδέσει την συμφωνία αυτή με μια βαθιά μεταρρύθμιση της υλοτομίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας προϊόντων ξυλίας είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την ικανότητα της συγκεκριμένης χώρας και της συγκεκριμένης κυβέρνησης να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να έχει την πολιτική βούληση για να το κάνει. Ιστορικά θα έλεγα ότι η συμφωνία με την Ινδονησία είναι το παράδειγμα στα πλαίσια του οποίου η διαπραγματευτική διαδικασία συνοδεύθηκε θα έλεγα ε, για να μην πω ότι ακολούθησε τις διαρθρωτικές αλλαγές στον τομέα της παραγωγής και επεξεργασίας ξύλου. Τώρα, για κάποιες εσωτερικού τύπου εμπορικές δραστηριότητες μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις και αποκλήσεις. Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο βασικός στόχος αυτών των εθελοντικού τύπου συμφωνιών είναι πάντα καρπός ε, διαπραγματεύσεων. Οι εταιρικέ συμφωνίες από τη μία και οι εθελοντικές συμφωνίες από την άλλη έχουν σαν βασικό στόχο την ενίσχυση του διαλόγου ανάμεσα ε, στην βιομηχανία, την συγκεκριμένη και την κοινωνία των πολιτών. Ευχαριστούμε. Ε, νομίζω ότι βασικά έχουμε τον ίδιο στόχο, έχουμε ένα κοινό όραμα αν θέλετε και όλοι συμφωνούμε ότι το VPA αυτό θα πρέπει η εθελοντική αυτή συμφωνία να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί το ταχύτερο δυνατόν όπως είπε και ο κύριος Ζαχράντιλ θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε, πριν από την επικύρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιετνάμ. Ένα από τα σημαντικά θέματα στα πλαίσια της συμφωνίας είναι ε, η συζήτηση για την αηφόρο ανάπτυξη. Το κείμενο αναφέρεται σε δύο δεσμευτικά μέσα, το Ε, υπάρχει δηλαδή αναφορά και σε σχέση με τα θέματα της ε, νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας και σε σχέση ειδικότερα με τα προϊόντα αλίας και ιδιαίτερα με τα προϊόντα παράνομης αλίας. Το να περιλαμβάνονται, εν πάση περιπτώσει, κεφάλαια για την αηφόρο ανάπτυξη στις συμφωνίες αυτές ε, ελευθέρου εμπορίου θα συμφωνήσω με τον κύριο Προύστο ότι μια ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου δεν είναι ένας αυτός σκοπός. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει σαν ε, στόχο την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα συν ε, φυσικά αναγνωρίζουμε εδώ και την αηφορία. θα ήταν θετικό περισσότερο στι ασιατικέ χώρες να ακολουθήσουν την διαδικασία των εθελοντικού τύπου συμφωνιών. Άκουσα όμως ότι δυστυχώς μόνο η Μαλαισία, εκτός από την Ινδονησία και το Βιετνάμ, είναι διατεθειμένη και έχει προετοιμαστεί έτσι ώστε να συνάψει μια τέτοια συμφωνία. Χθε είχα την τύχη να συναντηθώ με τον Υπουργό Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Μαλαισίας και του είπα ότι η Μαλαισία πράγματι είναι πλήρως προετοιμασμένη να συνάψει μια τέτοια εθελοντική συμφωνία αλλά υπάρχει το θέμα μίας από τις συστατικές πολιτείες της Μαλαισίας, του Σαραβάκ, που δεν έχει ακόμα θέση σε λειτουργία α, α, τις αλλαγές αυτές. Και υπάρχει ισχυρά αποκεντρωμένη διοίκηση σε σχέση με τέτοια θέματα, πάντως ελπίζουμε ότι η Μαλαισία θα υπογράψει μια τέτοια συμφωνία με την Ένωση. Τώρα για το δικό σας ερώτημα κύριε Πρόεδρε, για το τι γίνεται σε σχέση με τον τομέα επεξεργασίας προϊόντων ξυλίας στο εσωτερικό της χώρας. Μετά την επίσκεψή μου στο Βιετνάμ πρώτα το 2013 και τότε ήμουν υπουργό για τη Διεθνή Ανάπτυξη, παρατήρησα ότι η Φιλανδία είχε υποστηρίξει μια καταγραφή του δασικού πλούτου του Βιετνάμ. Η προσπάθεια αυτή τώρα ολοκληρώθηκε, τώρα καρποφόρησε. Υπάρχει ένα open database, μια ανοιχτή βάση δεδομένων που λέγεται FOMIS, που ξεκίνησε από φιλανδική πρωτοβουλία είναι προσβάσιμη σε πολλούς ενδιαφερομένους, σε πολλές κατηγορίες εμπλεκομένων και ενδιαφερομένων γύρω από τα θέματα των δασικών πόρων. Αν έχει κανείς μια ανοιχτή πρόσβαση σε τέτοιου είδους βάσεις δεδομένων, μπορεί να δει κανείς αν ένα δάσος εξαφανίζεται, αν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι, και υπάρχει και ένα ερευνητικό κέντρο το οποίο παράγει ε, δορυφορικές φωτογραφίσεις κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σχετικά με τον έλεγχο της κάλυψης και τις πιθανές παράνομες υλοτομικές δραστηριότητες. Είναι λοιπόν αυτός ίσως ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε εφόσον διατηρήσουμε την δασική κάλυψη να συνεχίσουμε την αυξημένη απορρόφηση διοξιδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε ένα τέτοιο μέσο στη διάθεσή μας και θα πρέπει να το φροντίσουμε κατά κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι λοιπόν 25 Φεβρουαρίου. Πέμπτη απογευματινή. Και 18 ή 19 θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το θέμα υπαρίθμ 9. Είχαμε ήδη την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φιέλνερ. Και τώρα πλέον είναι καθήκον του Κρίστοφ να μας δώσει τη δική του άποψη για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τις τροπολογίες. Προς έκπληξή μου ήταν ταυτόσιμες όλες οι τροπολογίε δεν ξέρω ποιε είναι οι σκοτεινέ δυνάμει που οδηγούν στο αποτέλεσμα. Αυτό λέει ο μιλητή, αλλά έτσι ήταν. Υπάρχει μια γενική υποστήριξη προς το σύστημα, μερικές φορές όμως πρέπει να συζητούμε και για την υλοποιησιμότητα κάποιων από τις πιο καλές ιδέες, μεταξύ των οποίων είναι να προσθέσουμε και τη Συμφωνία των Παρισίων στη σύμβαση. Αλλά μιλώντας για υλοποιησιμότητα, ο μηχανισμός ε, ε, επισήμων καταγγελιών για την κοινωνία των πολιτών αυτό πρέπει να συνδεθεί με την συνεχιζόμενη παρακολούθηση. Γιατί διαβάζοντάς το, έχω την εντύπωση μερικές φορές είναι ότι θα ήθελα να αντικατασταθεί ο ILO από την επιβολή, από την παρακολούθηση και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η σωστή προσέγγιση. Εν πάση μπορούμε να συζητήσουμε και για το πώς θα λειτουργούσαν στην πράξη όλα αυτά. Γιατί για κάποιες από τις χώρες δικαιούχους όπως η Καμπότζη αυτό θα σήμαινε σημαντικούς πόρους και δέσμευση που συνήθως κάνουν μόνο μέσω FTA. Για την διαφάνεια είναι <clears throat> ένα θετικό στοιχείο αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο με τις χώρες αυτές και μόνο μέσω ειλικρινούς διαλόγου μπορούμε να συζητήσουμε για κάποιο είδου ε, περιθώριο ελιγμών για, τις, ε, για την ε, μεταποίηση των εξαγωγών. Αυτό αφορά σε περιφέρειες των ε, δικαιούχων χωρών και θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες προϋποθέσεις όπως και άλλες χώρες. Επίσης πρέπει να δούμε τι μπορούμε να τοποθετήσουμε Ε, προς την κατεύθυνση της ε, πληρέστερης και πιο αποτελεσματικής παρακολούθησης γιατί μερικές από τις χώρες αυτές εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο περιφερειακά και επομένω η πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν πολύ περιορισμένη στις χώρες αυτές. Υπάρχουν όμως και πολύ θετικές παρατηρήσεις πέραν της Συμφωνίας του Παρισίου αλλά και σημαντικές ε, διαφορές απόψεων. Εγώ νομίζω ότι το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για παράδειγμα οι Ηνωμένε Πολιτείε το βλέπουν ως ένα μέσο οικονομικού συμφέροντος. Δηλαδή η προτιμησιακή μεταχείριση ε, και το GSP Plus θα πρέπει να μείνει σε ένα σύστημα παροχής κινήτρων προς λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Και επομένω δεν συμφωνώ σε ένα γενικευμένο GSP σύστημα και ότι στην κατάργηση του μάλλον, γιατί αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο προς την γενική στόχευσή μας που είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας, της ένδυας. Πιστεύω πάντως ότι έχουμε μια καλή πιθανότητα να βρούμε συμβαστικές ε, λύσεις στις περισσότερες από τις τροπολογίες και προσβλέπω στην ε, συνεχιζόμενη συνεργασία μας ιδιαίτερα και εν των τροπολογιών Ντεβε και Ντροά. Ε, σας ευχαριστώ. Η Σκιώδης ε, S&D, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά, την ταχύτατη δουλειά, καθότι είχαμε και καθυστερημένη υποβολή της έκθεσης. Εμείς επιμείναμε ώστε να υποβληθεί το ψήφισμά μας γιατί θεωρούμε ότι το σύστημα ε, δεσμολογικών προτιμήσεων είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα που έχει η Επιτροπή προκειμένου να αναπτύξει τη σχέση της και να έχει σημαντικό αντίκτυπο μοχλό πίεση ε, με συγκεκριμένες χώρες. Η δουλειά αυτή είναι πολύ σημαντικά. σημαντική. Κάποιες από τις θεματικές που ανέφερε ο εισηγητής και για μας είναι πολύ σημαντικές και από αυτών τουλάχιστον θεωρούμε ότι μπορούμε να επιχειρήσουμε να έχουμε μια καλή συνεργασία, ενίσχυση της συμμετοχής ε, της κοινωνίας των πολιτών, ε, περισσότερη διαφάνεια, και καλύτερη επιτήρηση, παρακολούθηση. Ο λόγος τον οποίο εμείς υποβάλαμε τροπολογίες ήταν ακριβώς γιατί σε κάποια σημεία θεωρούμε ότι θα πρέπει να καταβληθεί μια περαιτέρω προσπάθεια. Υπό την έννοια ότι πρώτα απ' όλα θεωρούμε χρήσιμο να αναφερθούν ρητά περιπτώσεις κατά τις οποίες στην περίπτωση χωρών με τις οποίες έχουμε μία σχέση GSP αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και καθότι αυτό το μέσο είναι ένα μέσο ενίσχυσης, βοήθειας προς τις χώρες αυτές, ε, αντιστοίχως είναι και ένα μέτρο, ένα σύστημα δέσμευσης που θα πρέπει να αναλυφθεί από τις χώρες αυτές προκειμένου να βελτιώσουν και τα πρότυπά τους στο επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι και ο λόγος που επιμείναμε σε κάποιες τροπολογίες που θεωρούμε απολύτως υλοποιήσιμες και καθόλου ουτοπικές. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, μέσω των τροπολογιών που υποβάλαμε είναι μια σταδιακή βαθμία πρόοδος λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των χωρών αυτών αλλά δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι το γενικό μας σύνθημα δεν μπορεί να είναι η αξιοπιστία η οποία βασίζεται αφενός στην σαφήνεια των, του ποιε είναι οι αξίες μας και της διαβίβασης του μηνύματος αυτού προς τις χώρες αυτές αλλά και αφετέρου στο γεγονός ότι συνολικά η εμπορική, η εμπορική και η οικονομική υποδομή δεν μπορεί να υποστηριχθεί παρά μόνο εάν αποφύγουμε τους μηχανισμούς dumping κοινωνικού, περιβαλλοντικού, εργασιακού, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και που υποσκάπτει ε, την αξία των εμπορικών συναλλαγών αν θέλετε και στο ιστορικό της δικής μας αγοράς. Αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν συνοδεύσουμε το GSP με τέτοιες αξίες, αν δεν διέπουν αυτά το παγκόσμιο εμπόριο, τότε αυτό το σύστημα δεν θα μπορέσει να αντέξει στο χρόνο. Ο κύριος Κάρεμ δεν είναι εδώ. Η κυρία Ρίς για τους Άλντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, είναι η δική μου σειρά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο εισηγητή αναφέρθηκε σε κάποιες σκοτεινές δυνάμεις πίσω από τροπολογίε. Ε, εγώ εκ μέρου τη κυρία Λαλόν θα αναφερθώ σε κάποιες από αυτέ. Ε, και ελμίζω, ελπίζω δηλαδή ότι είμαστε από, από το καλό σύνορο ε, και όχι το κακό σύνορο αυτών των σκοτεινών δυνάμεων θεωρούμε ότι αυτό το σχέδιο ψηφίσματος είναι ε, θεμελιώδης σημασίας προκειμένου να υλοποιήσουμε ένα σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων που παραχωρούμε προς τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες που θεωρούμε ότι μπορεί να συνεισφέρει στην σταθερότητα την οικονομική και κοινωνική των δικαιούχων χωρών. Οι τροπολογίες της ε, κυρίας Λαλόντα στοχεύουν ακριβώς στην ανάπτυξη των ε, εμπορικών συναλλαγών εντό ενό πλαισίου που να είναι θετικό και ισορροπημένο. Η κυρία Λαλόντ υπέβαλε 7 τροπολογίες επί 5 αξώνων που τις φαίνονται ουσιαστική σημασία για την καλή λειτουργία του κανονισμού αυτού. Καταρχά, οι στόχοι βιωσίμου ανάπτυξη. Ε, πρέπει να χαίρουν περισσότερες προσοχές γιατί στο GSP Plus θα πρέπει να σεβόμαστε 27 θεμελιώδη σημασία σε διεθνείς συμβάσεις και μας φαίνεται πολύ σωστό να προσθεθεί και η Συμφωνία του Παρισίου. Δεύτερον, η παρακολούθηση των διεθνών αυτών δεσμεύσεων σημαίνει και το ανέφερε και η, η σκιώδης του SND την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών γιατί μόνο με τέτοια δέσμευση μπορούμε να ε, βοηθήσουμε να υποστηρίξουμε και τη δουλειά της δικαιοσύνης και των ομοδίων αρχών. Τρίτον, είναι σημαντικό να έχουμε στοχευμένη προσέγγιση που να ε, επωφελεί όχι μόνο κάποιες, κάποιους τομείς της οικονομίας, αλλά ένα, το ευρύτατο δυνατό φάσμα των ε, φορέων και εμπορικών εταίρων από του συμβαλωμένου. Επίσης η συμπερίληψη των υπηρεσιών στο GSP ε, φαίνεται στην κυρία Λαλόντ ίσως ε, υπερβολικά φιλόδοξη και ίσως και αντιπαραγωγική. Ε, έχουμε κάποιε αμφισημίες εδώ, θα θέλαμε λοιπόν να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο το σημερινό για να έχουμε απτές οικονομικές βελτιώσεις και συμπερασματικά τα κλώστο υφαντουργικά δεν υπάρχουν στο σχέδιο ε, που είναι όμως τομέας που υπερισχύει στις εισαγωγές ε, υπό το GSP και επομένως το σημείο 12 θα πρέπει να ανασ... αναδιατυπωθεί με περισσότερη σαφήνεια. Σας ευχαριστώ. Κύριος ε, Σάντι, Δεν είναι παρούσα η συνάδελφος, οπότε θα διαβάσω το έγγραφό της. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα στηρίξω κάποιες από τις τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν στο μέλλον την κατάσταση, αλλά υπάρχει ένα θέμα με ορισμένες τροπολογίες με την 81 για την εξαίρεση ορισμένων προγραμμάτων από τα GSP. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όμως κάποιες τέτοιες ζώνες, αλλά θα πρέπει να γίνει αυτό μέσω της εφαρμογής των τοπικών ρυθμίσεων που θα σέβονται τις διεθνείς συμφωνίες. Για τη σταδιακή τώρα ανάκληση δασμολογικών περιορισμών ε, η λογική λέει η συνάδελφος ότι ακολουθεί ε, όχι τη λογική της αιρεσιμότητας αλλά την απλή κατάργηση κάποιου τέτοιου τύπου δασμολογικών ε, Επίσης η επεξεργασία των παραπώνων και αναφορών στις συγκεκριμένες χώρες θα πρέπει να γίνεται από διαφορετικά επίπεδα Ελπίζω όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τελικά να κάνει μια πληρέστερη πρόταση. Και τέλος, τροπολογίες 122 ε, και 124 εκεί όπου θεωρείται ότι δεν είναι ανεπαρκή τα εθελοντικά σχήματα και συμφωνίες Ίσα ίσα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ιδιωτικά προγράμματα και στον τομέα της συμμόρφωσης. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η ανυπαρξία διακανονιστικού πλαισίου και νομικών ρυθμίσεων, το πρόβλημα είναι η επιβολή των ρυθμίσεων αυτών και ο έλεγχος. Αυτά λέει ο σκιώδης μας ο κύριος Καρίμ. Ευχαριστώ πολύ για την κυρία Μινέρ. Όπως είπα η Λόλα Σάντσες είναι ισκιώδης, δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα. Θα πρέπει, λέγει η κυρία Σάντσες, να, προσπαθήσουμε, να προσπαθήσουμε συγγνώμη, να δούμε ποιος είναι ο βασικός στόχος, η μείωση της φτώχειας. Όχι να περιοριστούμε σε σχέση με το ισοζύγιο το εμπορικό ή κάποιες άλλες τεχνικές και αριθμητικές ρυθμίσεις, αλλά να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής. Σεβόμενη την αηφορία, θα πρέπει επίσης ε, τα θέματα της παιδείας να ληφθούν υπόψη και το θέμα των κυρώσεων με την δυνατότητα επιμέρους απόσυρσης. Η αρμόδια επιτροπή υιοθέτησε τη δική της γνωμοδότηση χθες, ομόφωνα σχεδόν, και ελπίζω και αυτή η Επιτροπή να κάνει το ίδιο. Θα συνεχίσω τη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις έτσι ώστε να υπάρξει ε, σωστή αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει το θέμα της ανάπτυξης ε, στον τομέα της χωροταξίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υπονόμευσης των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτό θα δείξει επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν συγκεκριμένα επίπεδα εφαρμογής της αρχής της ε, της οφειλόμενης συμμόρφωσης από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για το ΙΕΝΕΦ, κυρία Ζαμέ κάποιες σκέψεις για ένα σύστημα το οποίο είναι υποσυζήτηση τώρα και το οποίο με εκπλήσει λίγο γιατί διαρωτώ γιατί είμαστε εδώ σήμερα για να εκφράζουμε τη λύπη μας για την έλλειψη ποικιλία αν θέλετε κάποιων οικονομικών δραστηριοτήτων που ωφελούνται από τις δασμολογικές συμφωνίες που έχουν φυσικά ε, σαν βασικό αρνητικό ε, αποτέλεσμα την υπερεξειδίκευση και την αποκλειστικά, αποκλειστική ενασχόληση με τις εξαγωγικές καλλιέργειες, κάτι το οποίο δεν δίνει κίνητρα στην εσωτερική αγορά, ενώ φυσικά οι, ε, οι καλλιέργειες οι οποίες καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες είναι πολύ πιο ωφέλιμες και δεν επιτρέπουν καταχρηστικές χρήσεις ε, της καλλιέργειας της γης και βοηθούν επίσης ε, την ένταξη ε, των χωρών, ε, των παραγωγών από τις των τρίτων χωρών σε, στα συστήματα του διεθνούς εμπορίου, το οποία όμως δεν λειτουργούν με ικανοποιητικό τρόπο και πολλές φορές στρεβλώνουν τις οικονομίες των μικρών χωρών και των Darling. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τα όσα είπε η Αλέσσα ω η συζητήτρια μα. Εγώ υπέβαλα μια σειρά από τροπολογίε γιατί έγιναν μια σειρά από αναφορέ σε ε, θέσει ε, που ήδη οθέτησε ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη μεταρρύθμιση του Γενικευμένου Συστήματο Υποτιμήσεων και δεν συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω έκθεση. Ωστόσο, αυτέ οι θέσει είναι χρήσιμε και επαναλαμβάνω εδώ ότι αυτό το σύστημα GSP Plus είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξάλληψη τη φτωχία και για την προώθηση τη ανάπτυξη, αλλά προωθεί επίσης ε, και την ε, κύρωση από άλλες ε, χώρες των διεθνών συμβάσεων και κατά τη συνέπεια την ανάληψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις. Άρα λοιπόν μια σειρά από ζητήματα όπως για παράδειγμα η ανάγκη πολύ σαφών ορισμών ως προς για παράδειγμα το, την συστηματική, τις συστηματικές υποχρεώσεις και ούτω καθεξής είναι ζητήματα ε, τα οποία θα πρέπει να ορίσει η Επιτροπή, για παράδειγμα, ω προ το τι είναι η σαφή ε, και η συστηματική παραβίαση. Τέτοιου είδου σαφεί ορισμοί είναι πολύ σημαντικοί για τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, προκειμένου να ελέγχουν το πώ ε, συμπεριφέρεται μια συγκεκριμένη χώρα αποδέκτη του GSP. Μετά θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η εμπορική μα πολιτική σε γενικέ γραμμέ. Δηλαδή, στι νέε μα συμφωνίε συμπεριλαμβάνουμε πάντοτε και την εταιρική ευθύνη και κατά συνέπεια στην μονομερή εμπορική πολιτική την οποία ασκούμε προ τα έξω, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα και αυτή την πτυχή. Δηλαδή και στο πλαίσιο ακριβώ του συστήματο GSP, ε, με αυτόν τον τρόπο ε, επιβάλλοντα την ε, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συμμόρφωση με τι διεθνεί συμβάσει σε ό,τι αφορά ακριβώ το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και του κανόνε σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Ένα τρίτο σημείο είναι η εφαρμογή ενό δεσμευτικού μηχανισμού μέσω του οποίου η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει για την προστασία των δικαιωμάτων θα μπορούν να θίγουν τις ανησυχίες τους. Ε, και αυτό το έχουμε αναφέρει ευθύ εξ αρχής ότι Υπάρχουν κάποιε ανησυχίε οι οποίε έχουν εκφραστεί ε, προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά ακριβώ την υλοποίηση του συστήματο GSP ε, από τι χώρε από τι οποίε προέρχονται αυτέ οι οργανώσει. Αυτή λοιπόν τη στιγμή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο μηχανισμό μέσω του οποίου να υποβάλλονται αυτές οι καταγγελίες ε, και να επηρεάζουν τη διαμόρφωση του συστήματος GSP. Άρα λοιπόν θεωρώ πως είναι ε, κάτι το σωστό, δεν θεωρώ πως είναι αδύνατο να εφαρμοστεί και δεν θεωρώ πως επιβάλλει υπερβολικά μεγάλο άχθος, δηλαδή το να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα επιτρέπει στις οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα να υποβάλλουν καταγγελίες. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα, θα είχαμε και μια πιο σφαιρική ε, αξιολόγηση των λόγων χωρών μέσω συστήματος οπόντο, μέσω scoreboard, ε, έτσι ώστε να ενισχύσουμε ακόμα, ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια. Τέλος, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν μια σειρά από χώρες οι οποίες ε, πέρασαν πλέον από το GSP Plus στην Συμφωνία σε Ελεύθερο εμπορίο ειδικότερα στη Λατινική Αμερική, όπου βέβαια σημειώνονται σημαντικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, και εγώ ενδιαφέρθηκα ιδιότερα κατά την δική μου βουλευτική θητεία στην ε, Γουατεμάλα και ε, την, τις εκτελέσεις εκεί που έγιναν για παράδειγμα και μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Άρα λοιπόν εκείνο που θα πρέπει να διασφαλίσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να μην έχουμε την περίπτωση όπου μεταβαίνουμε από ένα σύστημα GSP το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες υποχρεώσεις ε, που επιβάλλονται στα κράτη-μέλη σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μέσω των οποίων απαλλάσσονται από αυτές τις υποχρεώσεις ουσιαστικά. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν έχει αντίστοιχες υποχρεώσεις. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχουν τα κατάλληλα κεφάλαια ελοποίηση των συμφωνιών και διασφάλισης βιώσιμης ανάπτυξης από την πλευρά των λόγω χωρών. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρο. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω ε, μια συγκεκριμένη τροπολογία, την 126, η οποία ουσιαστικά ε, αποτελεί επανάληψη τη ίδια τροπολογία που είχε υποβληθεί σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση για την κλωστοϊφαντουργία και όπου αξιώνουμε να δίνεται προτεραιότητα, αν θέλετε, να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση για τα προϊόντα του fair trade, του δίκαιου εμπορίου. Ε, πάντοτε αναφερόμαστε στα ζητήματα παραβίασης ε, των υποχρεώσεων που απορρέουν από ορισμένε συμβάσει. Αλλά πάντοτε τα θύματα τέτοιου είδου παραβιάσεων είναι ε, οι άνθρωποι αυτών των χωρών, οι πολίτες αυτών των χωρών. Αλλά μια άλλη προσέγγιση σε σχέση με τον ελόγο μηχανισμό είναι ακριβώς να δώσουμε προτεραιότητα πρώτη μισιακή δηλαδή μεταχείριση σε συγκεκριμένα είδη προϊόντων όπως σε παράδειγμα του fair trade εφόσον πληρούν φυσικά ορισμένες προϋποθέσεις. Και πρόκειται δηλαδή για μια τροπολογία που τότε στην άλλη γνωμοδότηση είχε εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα να δώσω το λόγο στην Αλίνα Μπολκούχα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Χαιρετίζουμε αυτό το σχέδιο έκθεση από την πλευρά τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ και του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και παρακολουθήσαμε ε, στενά τις συζητήσεις ε, που γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο, χθε ειδικότερα στην ε, Επιτροπή ΑΦΕΤ. Κάτι δική μας άποψη, εν λόγω έκθεση, μας παρέχει πολύ σημαντικές, σημαντικά ρεθίσματα για σκέψη στο πλαίσιο του επόμενου GSP που θα αρχίσει να ε, ισχύει από τον επόμενο Ιανουάριο. Ε, είχαμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και σε εκείνη την έκθεση εξετάσαμε πιο συγκεκριμένα τρία στοιχεία, τρεις ε, στόχους ε, του GSP. Και επιχειρώ το γεγονό ότι αναφερθήκατε σε αυτά τα τρία στοιχεία εδώ στη συζήτηση. Το ένα από αυτά τα στοιχεία λοιπόν είναι μείωση τη φτώχεια και οικονομική ανάπτυξη. Το δεύτερο στοιχείο είναι βιώσιμη ανάπτυξη και η πρόθεση τη χρηστή διακυβέρνηση. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι η καλύτερη προάσπιση, η καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, με την βοήθεια λοιπόν ε, μιας εξωτερικής ε, επιχείρησης, ε, συμβούλου επιχειρήσεων, προβήκαμε σε αυτή την ενδιάμεση αναθεώρηση και διαπιστώσαμε ότι μέχρι στιγμής το GSP ανταποκρίνεται στους στόχους του, ειδικότερα στο πλαίσιο του προβλέψιμου πλαισίου που παρέχει στους ε, συμμετέχονται στις οικονομικές δραστηριότητες. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα σταθερό πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας για τα επόμενα 10 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, να πούμε ότι το GSP στο σύνολό του έχει παράσχει τεράστια πλέον εκτήματα για τις ευτοχότερες χώρες του κόσμου. Ειδικότερα στο πλαίσιο της προσέγγισης όλα εκτός από όπλο. Ε, και στο οποίο δηλαδή έχουν περιληφθεί όλες οι φτωχότερες ε, χώρες του κόσμου, 48 δηλαδή LDCs, με αύξηση κατά 62% του σχετικού Και οι χώρες που γενικότερα υποφελούνται από το ε, ε, σύστημα αυτό αύξησαν τη δραστηριότητά τους με μάσκα κατά 54%. Και αυτό δεν οφείλεται δηλαδή μόνο στην ε, στις εμπορικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά την εξαγωγική τους διαστηριότητα γιατί οι, αυτές οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,4% και το, από αυτές το 4,1% αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από εκεί και μετά εκείνο που προωθούμε ταυτόχρονα με το GSP είναι και διαφοροποίηση της παραγωγής και αναφέρεται και μέσα στην έκθεση δηλαδή πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτές τις χώρες έτσι ώστε να διαφοροποιήσουν τις εξαγωγές τους καθώς αυτή τη στιγμή τα τρόφιμα και ε, ο κλωστεφατουργικός τομέας είναι το οι οποίοι αποφελούνται ε, τα μάνα από το σύστημα GSP+. Αλλά υπάρχουν και άλλες ε, προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε, δηλαδή η, η αλυσίδα προμηθειών και ούτω καθεξής. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο το οποίο εξετάσαμε στην ανάλυση μας ήταν, όπως είπα, βιώσιμη ανάπτυξη και το κατά πόσο δηλαδή το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων διευκολύνει την κοινωνική ανάπτυξη, την προάσπιση των θεμελιωδικών εργασιακών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εδώ το συμπέρασμα της ε, μελέτης ήταν σαφές. Διαπιστώσαμε ότι ε, χάρη ε, στο monitoring, την παρακολούθηση την οποία προβαίνουμε και η οποία είναι πολύ εντατική και χάρη στις εκθέσεις που δημοσιεύουμε ένα-δύο χρόνια ασκούμε ισχυρές πιέσεις σε αυτές τις χώρες προκειμένου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις λόγω συμβάσεις απέναντι στους πολίτες τους. Αλλά ο εν λόγω θετικός αντίκτυπος δεν εξαρτάται μόνο από την προτιμησιακή μεταχείριση των λόγω χωρών. Εξαρτάται και το από το κατά πόσο ε, οι εν λόγω χώρε έχουν προβλέψει τι αντίστοιχε εμπορικέ πολιτικέ ούτω ώστε να υπάρχει και κατάλληλη διανομή ε, των ωφελών. Και Διαπιστώνουμε για παράδειγμα περιπτώσεις ε, φαρμακής εδαφών ή παραβίασης βασικών εργασιακών δικαιωμάτων σε ορισμένες χώρες. Και τρίτον, ένα τρίτο στοιχείο δηλαδή που ανέφερα ήταν ο αντίκτυπος αυτού του συστήματος ε, στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, στους ευρωπαϊκούς κλάδους. Ε, και αυτό σχετίζεται δηλαδή με το μηχανισμό διασφάλισης των συμφερόντων μας. Η χορήγηση λοιπόν των ελόγω προτιμήσεων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξήσει τις πιέσεις του ανταγωνισμού στις ε, ευρωπαϊκές βιομηχανίες και κατά συνέπεια μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το μηχανισμό ε, safeguard. Ε, για παράδειγμα, η αύξηση των ε, εισαγωγών από την Καμπότζη και το Μιανμάρ αποτέλεσε ένα πρόσφατο παράδειγμα ως προς την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Και επίσης υπάρχει και ένα σύστημα graduation, δηλαδή ένα σύστημα με βάση το οποίο υπάρχουν συγκεκριμένοι κλάδοι και συγκεκριμένες χώρες αποδέκτες του συστήματος που γίνονται υπερβολικά ανταγωνιστικές και κατά συνέπεια βγαίνουν από το σύστημα. Αυτό είναι λοιπόν σε γενικέ ε, γραμμέ το περιεχόμενο τη έκθεση ε, έχει προβεί σε συγκεκριμένε συστάσει. Ε, θα αναφέρω δύο. Αύξηση τη διαφάνεια και τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Άρα λοιπόν θα κάνουμε περαιτέρω προσπάθειε από την δική μα πλευρά για να διασφαλίσουμε ότι η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει, δηλαδή ζητείται η άποψή της πριν από παράδειγμα επισκέψεις για την αξιολόγηση από την δική μας πλευρά και η δεύτερη σύσταση σχετίζεται με την στενότερη εταιρική σχέση με τις εν λόγω χώρες. Δηλαδή πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη ευαισθητοποίηση του γενού σε αυτές τις χώρες αλλά και μέσω των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση αυτών των ε, προτιμήσεων. Άρα λοιπόν με βάση αυτές τις συστάσεις θα εργαστούμε μέσα στους επόμενους μήνες και από εκεί και μετά θα υπάρξει και μια αξιολόγηση αντικτύπου που θα λάβει ε, χώρα και η οποία θα λάβει υπόψη σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Γιατί η έκθεση στην οποία σας ε, αναφέρθηκα αφορούσε μια ε, περίοδο μόνο τριών ετών. Η επόμενη αξιολόγηση αντικτύπου αντιθέτω θα αφορά σε περίοδο έξι ετών. Ευχαριστώ, πρόεδρος, ο Κρίστοφ. Δύο παρατηρήσεις έχοντας ακούσει την συζήτηση αυτή και τις τροπολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη δομή του GSP. Γιατί συμφωνούμε, πιστεύω, όλοι για το γενικό στόχο της εξάλληψης της φτώχειας. Αλλά θεωρούμε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι πιο φτωχές χώρες στον κόσμο, θα πρέπει να λάβουν κάποια επιπλέον βοήθεια, κάποιο είδου επιπλέον βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Παρότι μπορεί να μην είναι οι καλύτεροι μαθητέ και έχουν προβλήματα. Είναι πολύ κακό να έχει κανείς ε, διαφθορά και καταπίεση, ακόμα χειρότερα όταν είναι και φτωχός. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χώρες με τις οποίες δεν έχουμε δυνατότητα μόχλευσης. Δεν έχουμε καρότα ώστε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιο είδους μαστίγιο για μια βελτίωση και των κοινωνικών τους ε, προστασιών, περιβαλλοντικών, θεμελιωδών δικαιωμάτων κτλ. στις πιο φτωχές χώρες από όλες χρειάζεται απλώς βοήθεια. Και αν συμφωνήσουμε σε αυτό το ουσιαστικό, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για τις τροπολογίες και να βρούμε ένα κοινό άξονα. Ιδάλλως θα πρέπει απλώς να σπαταλήσουμε πάρα πολύ χρόνο απλώς για να συνεννοηθούμε σχετικά με το τι σημαίνει ένα σύστημα GSP. Και ε, ε, πρέπει να θέσουμε ένα θέμα του τι ρόλο πιστεύουμε ότι διαδραματίζει η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Trade διεθνώς. Εμείς δεν θέλουμε να υποσκάψουμε το ρόλο των πολυμερών ε, ιδρυμάτων και φορέων, αλλά θέλουμε να τους υποστηρίξουμε επίπεδα και να τους χρησιμοποιήσουμε ως κεντρικό κομμάτι της προσπάθειάς μας παρακολούθησης. Γιατί όσο καλά και να είναι τα κίνητρά μας, οι προθέσεις μας, μάλλον, ε, διακινδυνεύουμε ε, λέγοντας ότι εμείς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα από, από σας, να υποσκάψουμε το κύρος αυτών των πολυμερών φορέων, των διεθνών αυτών φορέων. Νομίζω ότι με μια τέτοια προσέγγιση μπορούμε να βρούμε συνεννόηση και συνεργασία. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, καλή τύχη στην περαιτέρω συζήτησή σας με τους κοιόδες. 19 Φεβρουαρίου θα υποβληθεί η έκθεση. Έχουμε ένα μονόλεπτο διάλειμμα και μετά θα έχουμε τους συντονιστές. Ευχαριστώ.